Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, begrüße Sie alle zur weiteren Sitzung. Ich möchte darauf aufmerksam machen. Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε τη συνεδρίαση και θα ήθελα να πω ότι έχουν αλλάξει θέση τα σημεία 6 και τα σημεία 9 της ημερήσιας διάταξης. Ας αρχίσουμε λοιπόν την εξέταση των σημείων της ημερήσιας διάταξης με πειθαρχία, γιατί αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Είναι δύσκολα σαν που έχουμε την ημερήσια διάταξη και έχουμε και πολλούς και ενδιαφέροντες προσκεκλημένους. Ξεκινάμε με τον πρώτο προσκεκλημένο μας, εκπρόσωπο της Ουγγρικής Προεδρίας και χαιρετίζουμε τον κύριο Φέλεχη και τον ε, κύριο Νίτραγη. Ευχαριστούμε και τους δύο υπουργούς και τους καλωσορίζουμε. Ο κύριος Φέλεχη, Υπουργό Εθνική Ανάπτυξη, αρμόδιος για το κλίμα και την ενέργεια και ο κύριος Νίτραγη, Υφυπουργό Πληροφοριών και επικοινωνία. Ελπίζω να μην έκανα μεγάλο λάθος στην προφορά των ονομάτων σας. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας. Θα δώσω το λόγο στους υπουργούς να κάνουν παρέμβαση και μετά θα κάνουμε ερωτήσεις. Ξεκινάμε με σας. Ο κύριος Φέλικνη. Thank you very much. Before I switch to Ευχαριστώ πολύ και πριν αρχίσω να μιλώ ουγγρικά, θα ήθελα να σας, καταρχήν να σας καλησπερίσω. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ και θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας στην Επιτροπή σας. Θα σας παρουσιάσω τη δομή της κυβέρνησής μας και του Υπουργείου Εθνικής Ανάπτυξης για να σας εξηγήσω γιατί ήρθαμε και οι δύο εδώ για να παρουσιάσουμε τα θέματα που αφορούν την Επιτροπή σας. Μετά την κυβερνητική αλλαγή που είχαμε πριν από 7 μήνες, έχουμε νέα Υπουργεία και ένα από αυτά τα Υπουργεία αποκαλείται Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης και ασχολείται με διάφορα θέματα. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και παραδοσιακά θέματα υποδομών, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές, όπως επίσης και η πολιτική συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης και η διαχείριση των ε, κρατικών πόρων και των δημοσίων συμβάσεων. Ένα ε, Υπουργείο με πολλές αρμοδιότητες λοιπόν και ε, επειδή ως Υπουργείο είμαστε υπεύθυνοι για, διάφορα, για διάφορους σχηματισμούς του Συμβουλίου κατά την Ουγγρική Προεδρία. Κάναμε αυτό διαχωρισμό και ο Υφυπουργός κ. Νιτραγή είναι αρμόδιος για το τομέα των τηλεπικοινωνιών και εγώ ασχολούμαι με τα υπόλοιπα θέματα. Θα αρχίσω τώρα να μιλάω στα Ουγγρικά για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι βουλευτές, για μένα είναι μεγάλη τιμή να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας στον τομέα της ενέργειας. Είναι στόχος της Ουγγρικής Προεδρίας να δημιουργήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη και ελπίζουμε ότι θα δώσουμε τον αρμόζοντα ρόλο στην πολιτική ενέργεια στο πλαίσιο αυτής της φιλοδοξίας. Κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας θα ασχοληθούμε με διάφορα στρατηγικά έγγραφα. Θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε το μέλλον της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, καθώς και τα μέσα που θα μας χρειαστούν γι' αυτό η Ουγγρική Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια μέσα στο επόμενο εξάμεινο να... και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων υπάρχει η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και ο στοχος 2020 20 στον τομέα της ενέργειας. Η Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου έχει προγραμματίσει στις 4 Φεβρουαρίου ε, ένα συμβούλιο για θέματα ενέργειας ε, και θέλουμε να τονίσουμε το ρόλο της πολιτικής ενέργειας ως πυλώνα των ευρωπαϊκών πολιτικών και θα ασχοληθούμε με συγκεκριμένα ζητήματα και ελπίζουμε να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις που θα ανοίξουν το δρόμο για το μέλλον. Και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένα συμπεράσματα στην διάσκεψη κορυφής. Η προετοιμασία της ε, πολιτικής για την ενέργεια ξεκίνησε τα περασμένα χρόνια και υπάρχουν προτεραιότητες ε, μεσοπρόθεσμες στους τομείς ε, που μας ενδιαφέρουν. όπως η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η αποτελεσματικότητα της ενέργειας, οι υποδομές, καινοτομία και έρευνα η εθνική ενεργειακή πόρη και οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας. Η Προεδρία του Συμβουλίου θεωρεί ότι στις προαναφερθήσεις πρωτοβουλίες θα είναι χρήσιμο να έχουμε πολιτική συνεργασίας Και βέβαια οι προτεραιότητε αυτές χρειάζονται χρηματοδότηση είτε από εθνικές είτε από ευρωπαϊκές πηγές και εδώ θεωρώ χρήσιμο να τονίσουμε ότι θα πρέπει ε, να φροντίσουμε και εμείς και εσείς από πλευράς του Κοινοβουλίου να θεσπιστεί το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Έχουμε αυτές τις προτεραιότητες μέχρι το 2020 και θα συνεχίσουμε με την επιδίωξη των στόχων αυτών και ε, ακόμη περισσότερο μακροπρόθεσμα. Η στρατηγική αυτή για την ενέργεια ε, συμπεριλαμβάνει την δημιουργία υποδομών και θέλουμε να μειώνονται οι χρόνοι που είναι απαραίτητοι για τις ε, αδειοδοτήσεις για να προωθήσουμε τις ε, πολιτικές μας προτεραιότητες. Έτσι πιστεύουμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματική η ενεργειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί έναντι τρίτων χωρών όλοι οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται την ασφάλεια που παρέχει η ενεργειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική ενέργεια θα πρέπει επίσης ε, να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το έγγραφο αυτό έγινε πριν από τις εβδομάδες από το Συμβούλιο. Έχουμε προς το παρόν προσωρινές θέσεις και κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας θα ασχοληθούμε περαιτέρω με την εξέταση ε, του κειμένου που έχουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου και στην ε, διάσκεψη κορυφής για την ενέργεια το Φεβρουάριο. Θα προωθήσουμε τους στόχους ε, αυτούς σε συνδυασμό με τη στρατηγική για το 2020. Ε, θέλουμε να υπάρχει συνέπεια της πολιτικής ενέργειας ε, με τους στόχους που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως τους στόχους ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όπως επίσης και τους στόχους για τη μικρότερη κατανάλωση προϊόντων άνθρακα μέχρι το 2050. χρειάζεται δημιουργία έξυπνων δικτύων και προώθηση των δικτύων αυτών και θέλουμε όλο και περισσότεροι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες υποδομές. Οι στόχοι μας συμπεριλαμβάνουν και τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα και συνεργασίες με τρίτες χώρες. με τις κατάλληλες επενδύσεις για την προώθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σε συνδυασμό με την χρηματοδότηση θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι βασικές αρχές για τους καταναλωτές και τους χρήστες. Η Επιτροπή προωθεί επενδύσεις πάνω από 1.000 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020 που θα είναι απαραίτητα για τη δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει ε, να ε, καταλήξουμε στη συμφωνία για το πώς θα χρηματοδοτηθούν τα κατάλληλα προγράμματα, ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης, ποιοι διάδρομοι θα έχουν προτεραιότητα και ποια έργα θα υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα. Κατά το 2011, η Επιτροπή θα κάνει μία σύσταση για την χρηματοδότηση των ενεργειακών υποδομών και κατά την Ουγγρική Προεδρία θα γίνει μία διάσκεψη για τις υποδομές στον τομέα της ενέργειας και αυτό θα γίνει στις 16 και 17 Μαΐου. Το θέμα της ε, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της ενέργειας είναι άλλος ένας στόχος και αποτελεί και ένα από τους πυλώνες ε, της πολιτικής της ε, Ουγγρικής Προεδρίας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα στους επόμενους μήνες να θέσουμε το πλαίσιο που θα αποτελέσει τη βάση για τα μελλοντικά μας βήματα. Ε, θα ληφθούν υπόψη οι συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο και με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία ε, νομίζω ότι θα παραμείνει η ενεργειακή αποδοτικότητα ε, ως προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω το δυναμικό εξοικονόμησης πόρων από την ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. και ε, η, ανάπτυξη θα πρέπει να, η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να αποδεσμευθεί από τις πρόοδους στον τομέα της ε, ενέργειας. Η πολιτική αυτή θα έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές στην Ευρώπη που θα επιβαρυνθούν με μικρότερο κόστος για την κατανάλωση ενέργειας. Συνεργαζόμαστε επίσης και με άλλες χώρες που έχουν παρόμοια συμφέροντα όπως και εμείς όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και ε, οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο έχουν αποδώσει ιδιαίτερη σημασία και σε θέματα όπως ο οικολογικός σχεδιασμός και το οικολογικό σήμα που θα πρέπει να συνδυαστούν με πολιτικές σε άλλους τομείς όπως είναι οι κατασκευές και οι μεταφορές. οι δημόσιε συμβάσεις, οι επενδύσει ε, και η εκπαίδευση καθώς και οι ρυθμιστικέ διατάξεις είναι τομεί που πρέπει να ληφθούν υπόψη και προγράμματα όπως ε, το Smart Cities ε, θα έχουν επίσης προτεραιότητα κατά, τους, κατά τα προσεχή έτη. Με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής θα συνεχίσουμε εμείς ως Ουγγρική Προεδρία τις εργασίες προς την κατεύθυνση αυτή και με την με το Συμβούλιο του Ιουνίου ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Το Συμβούλιο, η Ουγγρική Προεδρία χαιρετίζει την προοπτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ενεργειακή πολιτική και την προοπτική μέχρι το 2050 και αυτός ο δικός χάρτης ελπίζουμε ότι θα είναι επιτυχημένος. Θα ληφθούν παράλληλα υπόψη, όπως είπαμε, οι προτεραιότητες για την Ευρώπη του 2020 και θα τονίσουμε την ακεραιότητα των ενεργειακών αγορών και τον κανονισμό για τη διαφάνεια στις ενεργειακές αγορές. Οι τελευταίες συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο κατέληξαν στο ότι χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά που θα σέβεται τα δικαιώματα των καταναλωτών και θα εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για την αγορά. Η διαφάνεια και οι σωστές πρακτικές θα έχουν μεγάλη σημασία και η Προεδρία του Συμβουλίου ε, θα προσπαθήσει, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Στις ε, αρμόδιες ομάδες εργασίες του Συμβουλίου ήδη έχουν αρχίσει σχετικές συζητήσεις και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε μια εικόνα για τη θέση του Συμβουλίου. Υπάρχουν ε, πολλά σημεία που είναι κοινά με την οδηγία MIFID και με άλλες ε, νομοθετικές διατάξεις. και θα συνεχίσουμε την ε, παράλληλη επεξεργασία των θεμάτων σε ε, πολλά συμβούλια. Και είμαστε ε, πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Θα προσπαθήσουμε που είναι δυνατόν να έχουμε συμφωνία σε ε, πρώτη ανάγνωση. Ούτως ή άλλως θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν και να έχουμε την πολιτική συμφωνία που θέλουμε και στην ε, ε, διάσκεψη του Ιουνίου. αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε μόνο σε συνεργασία με εσά και με τα κράτη-μέλη και γι' αυτό ελπίζω ότι θα υποστηρίξετε το πρόγραμμά μας. η Ουγγαρία ως μέλος των τριών ε, προεδριών ε, μετά την Ισπανία και το Βέλγιο συνεχίζει τις εργασίες των προηγούμενων ε, προεδριών και σε συνεργασία με την Πολωνία που θα έχει την επόμενη προεδρία θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια. Θα είμαστε ανοιχτοί για συνεργασία και για συμβιβαστικές λύσει. Σα ευχαριστώ πολύ και περιμένω τι ερωτήσει σα. Ευχαριστούμε πολύ και θα δώσω το λόγο στον κύριο Νίτραη. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι κυρίες και κύριοι, σας χαιρετίζω εκ μέρους της Ουγγρικής Προεδρίας και εκ μέρους όλων εκείνων που παρακολουθούν τη συνεδρίαση αυτή μέσω του διαδικτύου. Οι στόχοι της Ουγγρικής Προεδρίας είναι πολύ γνωστή η συνεργασία στην Ευρώπη, η στενότερη και βαθύτερη συνεργασία στην Ευρώπη πιστεύουμε ότι θα μας οδηγήσει σε μια ισχυρότερη Ευρώπη. Και νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Για τους συγκεκριμένους στόχους τώρα της Ουγγρικής Προεδρίας που όχι μόνο αυτούς που επίπτουν στη δική μου αρμοδιότητα, αλλά γενικότερα νομίζουμε ότι ε, και αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μόνο μετά από συνεργασία και διαβούλευση. Ε, μόνο ο διάλογος μπορεί να μας βοηθήσει και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι αν βασιστούμε στο διάλογο θα μπορέσουμε και πιο γρήγορα να προχωρήσουμε σε μια καινούργια Ευρώπη, ε, ένα καινούργιο κόσμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε την νέα Ευρώπη που ονειρευόμαστε όλοι για να μπορέσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε ε, εμείς. Σαν πρόεδρος του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών θα Έχω ελπίζω στενή ε, και αγαστή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως γινόταν και στο παρελθόν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μας βασίζεται ε, στην ε, ψηφιακή ατζέντα της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποφασίστηκε πέρσι και θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τη Βελγική Προεδρία για τις προσπάθειες που κατ κατέβαλα για το θέμα αυτό. Η ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό η Ουγγρική Προεδρία θέλει και αυτή να συμβάλλει για να εφαρμοστεί σωστά η ατζέντα αυτή. Ήδη ξεκινήσαμε ε, συμμετέχοντας στην πρώτη ε, ψηφιακή συνδιάσκεψη ξεκινώντας ένα διάλογο και συνεισφέροντας ε, όπως μπορούμε θα προωθήσουμε την ψηφιακή ατζέντα και με δύο νομοθετικές πράξεις. Η πρώτη θα σχετίζεται με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών. Είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών είτε ε, ασχολούνται με ε, την ψηφιακή τεχνολογία στη δουλειά τους είτε στο σπίτι τους. Ε, είναι γεγονός ότι είμαστε ευάλωτοι εάν δεν εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα θέμα αυτό. Η προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με την ενίσχυση της του καινούριου οργανισμού για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών ε, ότι πιστεύουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τα μελλοντικά μας βήματα. Χαίρομαι ιδιαίτερα ε, γιατί πραγματικά και στις συναντήσεις που είχα με τον κύριο Τσίτσεστερ, τον εισηγητή σας για συναφή θέματα, βλέπω να υπάρχει ε, ελπίδα για το μέλλον. Θα προσπαθήσουμε επίσης να εξασφαλίσουμε τις υποδομές, τις κρίσιμες υποδομές και γι' αυτό θα οργανώσουμε στην Ουγγαρία, στη Λίμνη Μπάλατον, μια συνάντηση των Υπουργών, θα λάβετε γνώση αυτού και η δεύτερη τώρα νομοθετική πράξη που θα προωθήσουμε είναι το ένα πρόγραμμα για τις, το φάσμα ραδιοφωνικών ε, συχνοτήτων πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορέσει να βοηθήσει μαζί βεβαίως και με την ψηφιακή ατζέντα στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Κομισιόν έχει κάνει ήδη σχετική πρόταση. Στις 6 Ιανουαρίου Ήδη για το θέμα αυτό ήδη από τις 6 Ιανουαρίου κάναμε ε, μια συνάντηση στη Βουδαπέστη ε, όπου έλαβαν μέρος όπου έλαβε μέρος η κυρία Κρούζ ο κύριος Χακμάρ και εγώ και συζητήσαμε τα βασικά ε, στοιχεία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για και εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τη Βελγική Προεδρία που ήδη δρομολόγησε τις εξελίξεις αυτές. Στις 3 Δεκεμβρίου έλαβα μέρος στην Υπουργική Σύνοδο που ασχολήθηκε με το ραδιοφωνικό φάσμα, με τις ραδιοσυχνότητες Ε, και τα συμπεράσματα της Συνόδου ε, αυτής είναι πολύ σημαντικά. Βλέπετε από αυτά ότι υπάρχει ε, ομοφωνία μεταξύ των Υπουργών ε, για κάποιες βασικές αρχές που βεβαίως και οι συζητήσεις βεβαίως θα πρέπει να συνεχιστούν. Η Ουγγρική Προεδρία θα προσπαθήσει να λάβει υπόψη της ε, υπόψη της, της απόψης όλων θα πρέπει να απαντήσει βασικά ερωτήματα βεβαίως ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά να συγκεράσει και τις απόψεις των διαφόρων κρατών μελών. Στη Γενέβη θα λάβει χώρο όπως ξέρετε όπου να είναι η συνδιάσκεψη σε σχετικά με τις ραδιοσυχνότητες σε διεθνές επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο και ε, την οποία βεβαίω θα παρακολουθήσουμε και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν υπόψη και εκεί τα συμφέροντα και οι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, η θεωρία όπως καταλαβαίνετε η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών και οι ραδιοσυχνότητες είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας. Απ' την άλλη περαιτέρω όμως μα, βεβαίως δεν θα αφήσουμε παραμελήσουμε και άλλες πρωτοβουλίες όπως την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το e-governance, η Κομισιόν θα δημοσιεύσει και την έκθεση για το roaming στην, στο εσωτερικό της Ευρώπης. Ε, θα πρέπει βεβαίως μέχρι τότε να συζητηθούν κάποια θέματα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μερικά βήματα μπροστά και για το θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, είναι είναι το θέμα το που σχετίζεται με την δορυφορική πλοήγηση και που έχει συζητηθεί επανειλημμένα και σε, διαφορετικά βήματα και βεβαίως αυτή τη στιγμή απασχολεί και διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 16 Ιανουαρίου η Κομισιόν παρουσίασε μια ανακοίνωση και ελπίζουμε ήδη το Μάρτιο να μπορούμε να το Συμβούλιο μάλλον μέχρι το Μάρτιο να έχει εξάγει συμπεράσματα τα οποία να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Βεβαίω οι εργασίε του Κοινοβουλίου και του κυρίου Κράμακ που ασχολείται με το που για το θέμα αυτό θα ληφθούν υπόψη. Ε, Παρακολουθούμε επίση τι εργασίε που γίνονται σχετικά με το Γαλιλαίο. Ξεκίνησε, Γαλιλαίο. Ξεκίνησε η Βελγική Προεδρία. συνεχίζουμε εμεί και ελπίζουμε παρόλο που είναι δύσκολο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να προσεγγίσουν οι απόψει των μεν τι απόψει των δε. Επίσης, ε, ε, κύριοι βουλευτές, οφείλω να πω ότι έχω μεγάλες προσδοκίες από τη συνεργασία μαζί σας και, έχω και, και περιμένω ότι η Ουγγρική Προεδρία θα μπορέσει να βοηθήσει να προωθηθούν όλοι θέματα τα οποία θα βοηθήσουν και τους πολίτες και ε, θα προωθήσουν πρωτοβουλίες δικές σας. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε στη διάθεσή μας ακόμα 25 λεπτά για να θέσουμε ερωτήσεις και να απαντηθούν οι ερωτήσεις αυτές. 13 συζήτησαν το λόγο, βρίσκονται ήδη στο κατάλογο των ομιλητών, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερη πειθαρχία στη διάρκεια αυτής της συζήτηση Σας παρακαλώ, ε, συγκεντρωθείτε και επικεντρωθείτε στην ουσία των πραγμάτων. Ο κύριος Γκούρκ είναι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να σας θέσω ένα θέμα, ένα ερώτημα σχετικά με την ε, ενεργειακή πολιτική. Με μεγάλη χαρά άκουσα ότι στις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας βρίσκεται η ενέργεια. Και βεβαίως υπάρχει οικονομική κρίση η οποία οποία, στην οποία αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο αλλά η ενέργεια δεν πρέπει που δεν είναι λόγο να παραμεληθεί. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτό λοιπόν που ε, τονίζει τη σημασία της ενεργειακής πολιτικής. Η υποδομή στον τομέα της ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί ε, χωρίς τις αναγκαίες υποδομές είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγηθούμε σε μια αποτελεσματική ενιαία αγορά. Υπάρχουν περιοχές, περιοχές στην νοτιοανατολική Ευρώπη ιδιαίτερα, οι οποίες έχουν πρόβλημα υποδομής, το είδαμε αυτό και σε σχέση με την... Ε, ε, με το φυσικό αέριο, χρειάζονται νέοι αγωγοί και νέοι πόροι. Γι' αυτό ρωτώ λοιπόν κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, πώς βλέπετε το μέλλον της, του προγράμματος Ναμπούκο, της δικτύωσης αν θέλετε, αν θέλετε βορρά-νότου. Ο κύριος Χέρτσοκ, η κυρία Χέρτσοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς. Ε, και ε, Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον ε, κύριο Υφυπουργό και για το έγγραφο που μας μοίρασε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις για τους τομείς στους οποίους εσείς είστε αρμόδιοι. Υπάρχουν θέματα με τα οποία συμφωνούμε και με τα οποία διαφωνούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, χαιρετίζω αυτά τα οποία μας είπατε. Να ρωτήσω κάτι που δεν αναφέρατε. Αλλά εγώ ως σκιώδης εισηγήτρια θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το σημείο και συγκεκριμένα τα πυρηνικά απόβλητα. Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Και η ερώτησή μου είναι πιστεύετε ότι ε, μπορείτε να βρείτε μια επίλυση του προβλήματος κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, αν και το Κοινοβούλιο ε, ε, καταθέσει ένα ψήφισμα προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, για την, τον ενεργειακό εφοδιασμό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και για το φυσικό αέριο. Ποια είναι η θέση σας. Ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και τους Υπουργούς και τους ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Ξέρουμε ότι είναι σε καλά χέρια η ενεργειακή πολιτική. Μιλήσατε για τις αγορές ενέργειας και για τη διαφάνεια στην αγορά ενέργειας. Ελπίζουμε ότι η Ουγγρική Προεδρία θα καταφέρει να κάνει ένα σημαντικό βήμα και θα δούμε πόσο μπορείτε να προχωρήσετε προς την κατεύθυνση που μας αναφέρατε. Στις 4 Φεβρουαρίου θα γίνει η διάσκεψη κορυφής για την ενέργεια. Πώς έχουν προχωρήσει οι εργασίες προς ε, τη διοργάνωση αυτής της διάσκεψης θα ασχοληθείτε και με την καινοτομία και την ενέργεια. Τι αποτελέσματα προσδοκάτε από αυτή τη διάσκεψη και ποιος είναι ο ρόλος τη Ουγγαρίας κατά τη γνώμη σα. Και άλλη μια ερώτηση προς τον Υφυπουργό κύριο Νίτραη. Αναφέρατε το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις και όλο και υψηλότερο κόστος εμπλέκεται. Ποια είναι η θέση της Ουγγαρίας για αυτό το θέμα. Ο κύριος ε, Μπατσιούτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές και θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς για την ενέργεια ε, θα αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι πολλά ε, ε, τα θετικά από αυτά τα οποία μας αναφέρατε για το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας. Θέλουμε να έχουμε ανεξαρτησία από εξωτερικούς ε, φορείς και από τις εισαγωγές από τέτοιες χώρες. και στο πρόγραμμά σας συμπεριλαμβάνεται και αυτή η πολιτική σε σχέση με τις εξωτερικές σχέσεις. Πώς θα διασφαλίσετε στο μέλλον ίσους όρους για, την, για τον εφοδιασμό σε ενέργεια. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμός των μέτρων και των δραστηριοτήτων μας Ακούμε όλο και συχνότερα ότι είναι πολύ σημαντικός ο συντονισμός για την ενεργειακή αγορά και για την προστασία από ε, επιθέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους δύο υπουργούς για την παρουσία τους. Λέω κύριο Σέντσιου. Η Ουγγρική Προεδρία είναι βέβαιη ότι θα μπορέσει να αναπτύξει μία μοναδική αποτελεσματική και αποδοτική πολιτική ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας της. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να δρά πολυμερός και όχι μονομερός ε, στα θέματα της ε, ενεργειακής ασφάλειας. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, διότι όπως αναφέρετε και εσείς στο πρόγραμμά σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται αυτή την πολιτική κατεπηγόντως. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Κύριε Ζαντό, ευχαριστώ κύριε Υπουργή. Κύριε Υπουργέ, για το κλίμα και την ενέργεια, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα υπάρξουν δύο πολύ σημαντικά σημεία. Το Συμβούλιο, το Εαρινό, θα μιλήσουμε ε, για το θέμα της μείωσης ε, των στόχων μας για το διοξίδιο του άνθρακος μέχρι το 2020. Το Κανκούν θα είναι σημαντικό για τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα και επομένως ε, αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να την τροφοδοτήσουμε αλλάζοντας τις φιλοδοξίες μας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύουμε ότι το 30% είναι θετικό για την Ευρώπη, όχι μόνο για τι διεθνεί διαπραγματεύσει, αλλά και για τα συμφέροντα των επιχειρήσεών μα και τη ανταγωνιστικότητά μα στην Ευρώπη. Πώ θα διεξαχθεί αυτή η συζήτηση στο Συμβούλιο από την Ουγγρική Προεδρία. Επίση, στι 4 Φεβρουαρίου, άλλη μια σημαντική στιγμή τη Ουγγρικής Προεδρία, είπατε πολύ σωστά ότι είναι προ όφελο όλων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμείνουμε για την εξοικονόμηση ενέργεια. Για τα τελικά συμπεράσματα του Συμβουλίου δεν βλέπω να υπάρχουν όμω πολλά πολλά μέτρα. Πολλά λόγια υπάρχουν, αλλά όχι συγκεκριμένα μέτρα. Νομίζετε ότι μπορείτε να έχετε κάποια φιλόδοξα μέτρα για τι ανακαινήσει κτηρίων, παραδείγματο χάρη. Κύριε Κολάρσκα ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερο που η Ουγγρική Προεδρία δίνει τόση σημασία στην ενέργεια. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Πολωνία και γι' αυτό είναι στενή η συνεργασία μαζί σας. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι ο στόχος της Προεδρίας σας είναι μια ισχυρότερη Ευρώπη. Αυτό που θα ήθελα να γνωρίζω είναι πώς ε, ε, θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη ε, στα πλαίσια της ενέργειας. Απαριθμίσατε τις προτεραιότητές σας, οι οποίες συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Αλλά πώς ε, θεωρείτε ότι μπορούμε να κάνουμε μια πιο ισχυρή Ευρώπη στα πλαίσια της ενέργειας. Σαφώς ένα στοιχείο είναι η κατασκευή υποδομών, αλλά δεν είναι μόνο στοιχείο, υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι επισέρχονται σε αυτή την περίπτωση. Στην Ευρώπη έχουμε περιτροπής προεδρία και έτσι φροντίζουμε να συνεχίζεται το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και ε, η κάθε προεδρία θέτει συγκεκριμένους και σαφείς στόχους. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποιος είναι ο σαφής στόχος της Ουγγαρίας στον τομέα της ενέργειας. Και ένα τρίτο σχόλιο, η ερώτηση αν θέλετε. Όταν συζητάμε υποδομές, Ακούμε διάφορες περιγραφές ή διάφορους περιγραφικούς όρους. Ακούμε η Κεντρική Ευρώπη, η Νότια Ευρώπη και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ή στη χρήση αυτών των όρων. Δεν θα ήθελα η Πολωνία να βρεθεί σε μια μαύρη τρύπα και να μην θεωρείται ούτε κεντρική ούτε νότια Ευρώπη. Σας παρακαλώ να το θυμάστε αυτό. Eh, eh, Ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς για τις παρουσιάσεις τους. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Η φιλοδοξία σας για τους ε, στόχους για το κλίμα. Εμείς στο Κοινοβούλιο συζητάμε για το κατά πόσο θα έπρεπε να περάσουμε σε ένα ποσοστό άνω του 20% για το 2020. Εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι μακροπρόθεσμα μέχρι το 2050 που παραδείγματα ή ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να αλλάξει ο στόχος τον οποίο έχουμε ήδη υιοθετήσει. Πρώτη ερώτηση αυτή. Δεύτερη ερώτηση. Η οτι θα πρεπει να φροντισουμε να αλλαξει ο στοχος τον οποιο εχουμε ηδη οθετησει πρωτη ερωτηση αυτη δευτερη ερωτηση η οδηγια για τα ραδιενεργά απόβλητα. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο θα συζητήσουμε στην Επιτροπή μας αύριο. Είμαστε στη διαδικασία διαβούλευσης και επομένως το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προτάσεις μας. Θα ήθελα να γνωρίζω τα εξής. Τι ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει η Ουγγαρία με την έγκριση αυτής της οδηγίας, δεν ανέφερατε κάτι και επίσης θα ήθελα να μου διασφαλίσετε κατά κάποιο τρόπο ότι θεωρείται ότι το Κοινοβούλιο είναι ισότιμο μέλος, λες και έχουμε μια διαδικασία συναπόφασης, διότι αυτό είναι θέμα δημοκρατίας για, την, για τον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Ευχαριστώ. Η κυρία Πιλάρτη Καστίγιο. Ευχαριστώ. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω τους Υπουργούς για την παρουσία τους. Ε, ευχαριστούμε την Ουγγρική Προεδρία που είναι εδώ σήμερα. Έχω μία πρόταση και μία ερώτηση. Η ερώτηση αφορά τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρονική επικοινωνία. Όπως είπε ο υπουργό, υπάρχουν δύο θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικά. Το ένα αναφέρεται στην οίκαια και το άλλο αναφέρεται ε, στο φάσμα. Όσον αφορά το φάσμα, θα ήθελα να γνωρίζω αν στις επαφές που είχατε μέχρι τώρα έχετε μια εικόνα της κατάστασης. Θεωρείτε ότι είναι πρόσφορο το έδαφος ώστε να προχωρήσει το θέμα αυτό σε πρώτη ανάγνωση, δηλαδή στη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Κατά την άποψή μου ε, είναι κατεπήγον το ζήτημα και θα έπρεπε ε, οι συμφωνίες για το φάσμα ε, και τα όσα έχει ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το παρόν να προχωρήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα για να μην καθυστερήσει η κοινωνία της πληροφορίας και να εφαρμόζεται η τεχνολογία το ταχύτερο δυνατόν για να μπορέσουμε να έχουμε και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Και για τον τομέα αυτό το φάσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου από αυτού. Δεύτερον, τον Ιούνιο ε, θα υπάρχει μία διάσκεψη για ψηφιακά θέματα που ετοιμάζεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να συμμετέχει και η Προεδρία και διαμέσου της Προεδρίας και το Συμβούλιο. Αυτή ήταν η πρότασή μου. Η κυρία Καρβάλιο. Ένα σχόλιο και μία ερώτηση για την ενεργειακή πολιτική. Το σχόλιο είναι ότι η έρευνα για την ενέργεια αλλά και η ανέπτυξη, η διάδοση, βέβαιων πρακτικών είναι πάρα πολύ σημαντική για την ενεργειακή πολιτική και δεν άκουσα αρκετά στις παρεμβάσεις σας και τις προτεραιότητες που μας αναφέρετε. Αυτό ήταν το σχολείο μου. Δεύτερον, μια ερώτηση οι πόλεις ε, ε, κάνουν πάνω από 75% κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη και αν θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές και να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των πόλεων αλλά με ολιστικό τρόπο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιοι είναι οι στόχοι της Ουγγρικής Προεδρίας. Ε, υπάρχουν κάποια προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πόλεις. Ε, σκοπεύετε να ενισχύσετε και να συνεχίσετε αυτά τα προγράμματα. Η κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τους ε, δύο υπουργού και εύχομαι κάθε επιτυχία στην ε, Ουγγρική Προεδρία. Έχω δύο σύνδημες ε, ερωτήσεις. Η πρώτη για τον Υπουργό Ενέργειας. Είπατε και πολύ σωστά ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων σας είναι η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Είναι ένα θέμα που το έθεσαν αρκετοί συνάδελφοι στι προηγούμενε παρεμβάσει του. Παραμένει ωστόσο γεγονό ότι ο στόχο τη ενεργειακή αποδοτικότητα το 20% μέχρι το 2020, δεν πρόκειται να επιτευχθεί και αυτό είναι κάτι που το αναγνώρισε ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα μιλώντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να σα ρωτήσω λοιπόν ποιε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε σκοπεύετε να πάρετε κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα και πολύ περισσότερο με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 4η Φεβρουαρίου για να υπάρξουν αυτά τα νέα δραστικά μέτρα και να καλυφθεί το χαμένο έδαφος προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και επίσης επειδή αναφερθήκατε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικότερα στο θέμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κύριε Υπουργέ έχει οθετήσει πρόσφατα ένα ψήφισμα με το οποίο ζητά να καταστεί δεσμευτικό ο στόχος της ενεργειακής αποδοτικότητας και ήθελα το σχολείο σας. Κύριε Σαντή ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Ουγγρική Προεδρία. Είστε μέρος των χωρών του Βίσραντ και μέρος του, της Τρόικας ας πούμε που ε, δημιούργησε η, συνθήκη της Λισαβόνας δε, μετά που σας έρχεται η Πολωνία πως ε, κοιτάζεστε ε, να εξελίσσονται τα πράγματα, για πείτε μας μερικά πράγματα. Και κάτι τι άλλο. Τι έχετε να μας πείτε για τις μελλοντικές σχέσεις με τους εμπορικούς μας εταίρους, αυτούς που θα έρθουν και ενδεχομένως στην Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή ε, εσωτερική αγορά ενέργειας. Επόμενο θέμα για τις επικοινωνίες. Ε, έχουμε τις οπτικές σύνες. Ε, έχουμε τους δορυφόρους. Ε, τι προκρίνεται από αυτές τις ε, τεχνολογίες εσείς. Ποια από αυτές τις τεχνολογίες προκρίνεται. Η κυρία Ρούσκο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό θέλε, τι συνέχεια θέλετε να δώσετε στη συνέχεια της Κανκούν. Ξέρουμε ότι η επόμενη σύνοδος ε, θα γίνει στον Τουρμπάν και θα είναι αποφασιστική σημασίας διότι εκπνέει ε, η συνθήκη του Κιώτο και δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση για να συνεχιστεί το Κιώτο. μπορείτε ήδη να κάνετε κάτι στη διάρκεια του εξαμήνου ώστε να αποτελέσει επιτυχές, ε, ε, να είναι επιτυχή συγγνώμη, αυτή η σύνοδος ε, στον Τούρπαν. Θα ήθελα τώρα να στραφώ στον άλλο υπουργό και θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ένα τμήμα του φάσματος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και ενίσχυση δημοσίων υπηρεσιών μη εμπορικών στην Ευρώπη. Κύριε Τχοντμάν, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μια ερώτηση προς τον Υπουργό Τηλεπικοινωνιών. Η επιτυχία του προγράμματος της Προεδρίας σας εξαρτάται κατά πολύ από την συμφωνία που μπορεί να βρεθεί μέσα στο Συμβούλιο και υπάρχουν δύο είδη χωρών, όπω είδαμε και από το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Οι χώρε που έχουν προχωρήσει πολύ στην απελευθέρωση των υπηρεσιών και στη βέλτιστη χρησιμοποίηση του φάσματο, όπω η Σουηδία, παραδείγματο χάρη, και χώρε ε, που ε, είναι περισσότερο προστατευτικέ σε σχέση με μια κοινή στρατηγική. Πώς θα ε, μπορέσετε να μειώσετε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο τύπων χωρών. Δεύτερον, ε, υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ των διαφόρων εταίρων, αυτών που ε, παρέχουν προγράμματα, των ε, διαχειριστών του δικτύου κλπ. για την αποτελεσματικότητα του φάσματος. Έχουμε ζητήσει τη γνώμη και της Επιτροπής και θα ήθελα να γνωρίζω τη γνώμη της Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ, Λε Πρόεδρο. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από του υπουργού να απαντήσουν. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, το συντομότερο δυνατόν όμω θα θέλαμε τι απαντήσει σα. Ο κύριο Φέλιχη λίγα λεπτά έχετε στην διάθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μου αφήνει δύο λεπτά χρόνο ο Πρόεδρος για τις απαντήσεις μου. Θα προσπαθήσω λοιπόν. Εγώ θα είχα ζητήσει τρία λεπτά. Δεν είναι δυνατόν να απαντήσει κανείς διεξοδικά όλες τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω όμως ε, ε, να δώσω απαντήσεις και σας υπόσχομαι για κάποια ερωτήματα να σας στείλω και γραπτός απαντήσεις. Και αν θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο να γίνει μια σχετική συζήτηση και εγώ και ο συναδελφός μου θα είμαστε στη διάθεσή σας ε, άλλη φορά για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, πολύ συνοπτικά θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις απαντήσεις μου, όχι τις ερωτήσεις με τη σειρά δηλαδή, αλλά να απαντήσω δίνοντας μια συνολική απάντηση. Νομίζω ότι μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας είναι η πολιτική της ενέργειας σε συνδυασμό με την πολιτική για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό στον τομέα της πολιτικής για την προστασία του κλίματος ε, να συγκεντρώσουμε πολλούς εμπειρογνώμονες ε, οι οποίοι θα προετοιμάσουν και τη διάσκεψη κορυφής ε, στη Νότιο Αφρική για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή θέση και να μπορέσουμε να εκφραστούμε με μια κοινή φωνή στην Νότιο Αφρική. Κάναμε πολλά βήματα στην ε, διάσκεψη στο Κανκούν και πιστεύω ότι ήταν ε, επιτυχημένη ε, σε πολλούς τομείς. Δεν επέτυχε όμως ένα τομέα στην παράταση του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Εδώ είναι μια δέσμη μέτρων στην οποία πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα και θα πρέπει η ενέργεια και το κλίμα να προχωρήσουν με συνδυαστικά μέτρα και να διατυπώσουμε τις κατάλληλες προτάσεις ε, για την προστασία του κλίματος, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για χώρες εκτός Ευρώπης και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι χώρες υψηλών εκπομπών συνήθως. και μεταξύ των κρατών μελών ε, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το 20-30% όχι μόνο στο Κοινοβούλιο αλλά και μέσα στα κράτη-μέλη γενικότερα. Υπάρχουν ε, διαφορές απόψεων για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Και στον τομέα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος, ε, τα κράτη-μέλη δείχνουν ότι έχουν μια προθυμία να καταλήξουμε σε συνένεση αλλά δεν υπάρχει συνένεση για, για δεσμευτικούς στόχους. Η Ουγγρική Προεδρία θα συνεχίσει την ανταλλαγή απόψεων και θα προσπαθήσουμε να παραδώσουμε τη σκητάλη στην Πολωνική Προεδρία έχοντας κάνει ό,τι μπορούμε καλύτερα για να επιτύχουν εκείνοι ίσως πιο συγκεκριμένους στόχους. σε συνεργασία με την Επιτροπή και για το έγγραφο το οποίο προετοιμάζεται ε, για το Φεβρουάριο. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε μια ενιαία ενεργειακή ε, πολιτική. και θα προωθήσουμε την ανάπτυξη υποδομών διαφάνεια στη αγορά ενέργειας και επίτευξη ενός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου. Αυτά είναι στοιχεία που είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή πολιτική και όχι κατακαιρματισμένη πολιτική. Η διαφοροποίηση ε, των πηγών και των δικτύων είναι επίσης ένας στόχος για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ανεξαρτησία στον εφοδιασμό ενέργειας. Αναφέρθηκε το Ναμπούκο, υπάρχουν λύσεις όπως το Ναμπούκο, ΣΥΝ και άλλες λύσεις, το διάδρομη ε, βορρά-νότου. Όλες αυτές είναι κατευθύνσεις που θα καθορίσουν τις μελλοντικές μας πολιτικές για να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού σε υψηλό επίπεδο. Όντως δεν ανέφερα στην παρουσίασή μου τα ραδιενεργά απόβλητα. Κατά τη φάση προετοιμασίας δεν είχαμε τα σχετικά έγγραφα, τα λάβαμε αργότερα. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την ε, έκθεση αυτή εγκαίρως, νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο να προχωρήσουμε. Και θα προσπαθήσουμε να ε, προχωρήσουμε στη διαδικασία αυτή για να είναι ε, σε κατάλληλο στάδιο και να τη συνεχίσει και η Πολωνική Προεδρία. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνονται αυτέ οι διακρίσει βορρα βορρά-νότου η ανατολή ανατολή-δύση για τα ενεργειακά δίκτυα. όντω, ε, σωστά αναφέρθηκε για την Πολωνία και για τις ομάδες του Βίζεγκρατ. Χθε ήμουν στη Βρατισλάβα ε, σε μια συνεδρίαση και συζητήσαμε για την κοινή ενεργειακή πολιτική και τις ενεργειακέ ε, υποδομές και για του στόχους που θέτουμε ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα για την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις κατευθύνσεις της ενεργειακής ε, πολιτικής. Ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε ε, σημαντικές προόδους. η συνεδρίαση του Συμβουλίου που θα ασχοληθεί με τα θέματα της ενέργειας ως δεύτερο θέμα έχει το θέμα της καινοτομίας γιατί δεν, να, δεν μπορούμε να έχουμε σωστή ενεργειακή πολιτική χωρίς σωστή τεχνολογία και καινοτομία. Αυτά από μένα για τις απαντήσεις μου και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου για τις υπόλοιπες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να επικεντρώσω τις απαντήσεις μου στα σημαντικότερα θέματα. Βεβαίως όλες οι, οι ερωτήσεις ήταν ενδιαφέρουσες. Κύριε Μεσαρός, η, το ερώτημα που θέσατε ε, έχει στρατηγικές διαστάσεις. Το πρόγραμμα καλλιλέο είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, όλοι. Ε, τελικά οι Αμερικάνοι έχουν το GPS, οι Κινέζοι έχουν δικό τους σύστημα και οι Ευρωπαίοι χρειάζονται και αυτοί ένα σύστημα. Πρέπει να αφιερωθούν πόροι. Ε, για, να, για την εξέλιξη του συστήματος αυτού. Όμως α, οι πόροι αυτοί θα υπάρχουν από το 2016 και μετά. Μέχρι τότε δεν χρειάζεται να... Α, ε, δεν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Τώρα, ε, κυρία, κυρία μου, έχουμε ήδη συζητήσει μαζί ε, το σύστημα GNSS πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα, πρόγραμμα εδώ ε, και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ασχολείται με το θέμα αυτό. Εγώ οργανώνω τις ε, συνεδριάσεις αυτές και σε σχέση με την ψηφιακή ατζέντα θα θέλαμε να οργανώσουμε μια πρώτη συνάντηση πολύ γρήγορα για να μπορέσουμε να ε, ξεκινήσουμε κάποια μέτρα. Κυρία Τρότμαν, έχουμε συζητήσει επανειλημμένα το θέμα μαζί νομίζω, το θέμα που θέσατε. Συμφωνούμε και συζητούμε συνεχώς ε, για την εφαρμογή του πακέτου των τηλεπικοινωνιών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι υπάρχουν διαφωνίες. Η ψηφιακή ενιαία αγορά με τις νέες τεχνολογίες της είναι κάτι που όλοι θέλουμε να εφαρμόσουμε. Εμείς βεβαίως υποστηρίζουμε την ουδετερότητα των τεχνολογιών Ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις πάντως και όπως είπε ήδη και ο κύριος Φέλγη ε, είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε άλλες ερωτήσεις είτε τηλεφωνικά είτε με email και προσδοκούμε ένα ενεργό διάλογο με σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ τους υπουργού. Ήδη χαιρόμαστε για τη συζήτηση που έγινε. Ε, πολλοί από εμά έχουν πάει βεβαίω στην Ουγγαρία και έχουν συζητήσει τη, το πρόγραμμα της Ουγγλικής Προεδρίας. Αυτή ήταν άλλη μια συζήτηση που βοήθησε ιδιαίτερα νομίζω.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 Πρέπει να προσέξουμε γιατί περνώντα από το ένα θέμα στη μερισία διάθεση να χάνουμε 5-10 λεπτά κάθε φορά. Σας ε, καλωσορίζουμε Κύριε Επίτροπε Έτιγκερ, έχετε ξανάρθει στην Επιτροπή μας. Δεν θα κάνω μια τεράστια εισαγωγή γιατί δεν έχουμε τόσο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Έτιγκερ. Παρακαλώ. Λοιπόν, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριοι βουλευτές, θα συνεχίσω ουσιαστικά κάποιο ε, χωρί το θέμα το, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Φλέγκη γιατί συνεργαζόμαστε ήδη από τον Οκτώβριο με την Ουγγρική κυβέρνηση για την, ε, ε, τα θέματα της ενέργειας και είμαστε σε επαφή και με την Πολωνική Προεδρία η οποία θα συνεχίσει το έργο της Ουγγρικής Προεδρίας. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι υπεύθυνο για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική αν θέλετε τα κράτη, εσείς είστε υπεύθυνοι τα κράτη-μέλη υπεύθυνα, αλλά σε πάρα πολλές ε, συζητήσεις και με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Ρομπάη και βεβαίως ε, με άλλους ε, υπεύθυνους από διάφορες κυβερνήσεις συζητήθηκα, συζητούνται θέμα ενέργειας και, με το, και η Επιτροπή, ο κ. Μπαρόζο και η, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησαν το συζητούν θέματα ενέργειας και έτσι το, η ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου θα είναι θέμα προτεραιότητας δυόμιση ώρες συζήτηση για τα συναφή θέματα να σας πω ποια είναι τα σημαντικά θέματα για μας. Πρώτον, αποτελεσματικό... ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Θα κάνουμε μια πρόταση για ένα σχέδιο δράσης για την αύξηση της, αποτελεσματικότητας, της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Θα σας το υποβάλουμε και εσάς βεβαίως και θα, εκεί θα μιλάμε και για το τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον και τι είδους εθνικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερο, θα υποβάλουμε μια ενδιάμεση έκθεση ως το δυνατόν πιο ψυχρή και αντικειμενική για την εσωτερική αγορά ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο βεβαίως, τι γίνεται στην εσωτερική αγορά, τι γίνεται κατά ο καταναλωτή, πώς προχωράνε τα πράγματα, αν υπάρχουν ε, προβλήματα νομικά, τεχνικά, ε, προβλήματα παρακολούθησης και εποπτείας και θα αναφερθούμε στο ότι πρέπει να επιταχύνουμε κάπως τα πράγματα γιατί το τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί και αυτό από το Μάρτιο. Ωστόσο, πολλά πράγματα δεν έχουν γίνει σε πολλές χώρες. Κύριο μεγάλο βάρος θα δώσουμε στην υποδομή τι χρειάζεται από άποψη κεντρικού αν θέλετε κοινού προγραμματισμού ε, τι χρηματοδότηση χρειάζεται ποιοι είναι φορείς χρηματοδότησης και τι γίνεται με την αδειοδότηση και τι και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε την εφαρμογή με γρηγορότερο ρυθμό, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε ε, δυναμικά ή αν θέλετε άλλου είδους εμπόδια ε, για να επιταχυνθεί η δημιουργία υποδομών που είναι απαραίτητες. Θα αναφερθούμε επίσης στο θέμα της έρευνας στον ενεργειακό τομέα και θα προσπαθήσουμε να ε, να κάνουμε μια κάποια διαφήμιση αν θέλετε ούτως ώστε να διοχετευθούν περισσότερα κονδύλια από τον προϋπολογισμό για θέματα ενέργειας όπως το ΙΤΕΡ και τα Και θα, τέλος θα αναφερθούμε και στο Smart Cities and Communities έχουμε κάποια προγράμματα φάρους, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, για το θέμα αυτό. Αυτά, αυτές είναι οι βασικές μας προτεραιότητες που συναρθρώνονται πολύ καλά με την ενεργειακή πολιτική την οποία γνωρίζετε. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν θα πρέπει να συζητήσει αυτά και να φροντίσει να προωθήσει αν θέλετε τα θέματα αυτά και αυτό σαν ένα πρώτο βήμα για τον εξευρωπαϊσμό αν μπορώ να το πω έτσι της ενεργειακής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε που μας δίνετε και το χρόνο να θέσουμε ερωτήσεις και να ζητήσουμε απαντήσεις από εσά. Λοιπόν, αρχίζουμε τον κύριο Παλτσίτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για ε, την εργασία που έχετε καταβάλει μέχρι τώρα για τη δημιουργία της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας έχουν ήδη γίνει πολλά, αλλά ακόμη είναι πολλά αυτά τα οποία απομένουν να γίνουν για να μπορέσει η Ευρώπη να έχει ενεργειακή ασφάλεια. Ελπίζω λοιπόν ότι θα προωθήσετε τις ιδέες προς αυτή την κατεύθυνση. και ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και σε τοπικό επίπεδο τα οποία πρέπει να επιληθούν. Θα πρέπει να τεθεί μια προθεσμία, ούτως ώστε να επιληθούν αυτά τα προβλήματα μέχρι τότε για τις υποδομές ε, και για να δοθεί η πολιτική όθηση για να προχωρήσουν τα σημαντικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάλληλη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. κύριε κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, για την οδηγία ε, για το νερό ε, θα πρέπει να προσέξουμε να μην παραμελήσουμε την ενεργειακή πολιτική και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμη θα ήθελα να πω ότι ε, στη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα μόνο στα όριμα προγράμματα και θα πρέπει να υποχρεώσουμε τις αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη να προωθήσουν ε, μόνο πραγματικά όρημα προγράμματα τα οποία θα μπορούν να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Και τρίτον, ε, σχετικά με το διοξίδιο του άνθρακος, Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να προωθήσουμε τους στόχους μας ε, μαζί με την ε, έξυπνη ενέργεια και τις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και εσάς για άλλη μια φορά κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ. ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε συχνά στην Ευρώπη είναι η έλλειψη επαρκούς συνέργειας ανάμεσα σε διαφορετικές στρατηγικής σημασίας πολιτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερθήκατε και αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό. Ε, μιλώντας για την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θέσατε ως πρώτο θέμα την πρόθεση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Είπατε ότι θα παρουσιάσετε ένα νέο σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα ε, που θα πρέπει να ληφθούν στο εθνικό επίπεδο. Και μιλήσατε μετά ε, για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, την πορεία εφαρμογής του δεύτερου και του τρίτου ενεργειακού πακέτου. Ένα από τα ζητήματα, κύριε Επίτροπε, ε, καθοριστικής σημασίας για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ιδιαίτερα στο δεύτερο ενεργειακό πακέτο, ε, είναι και τα τιμολόγια. Τα τιμολόγια, τα οποία με βάση την Οδηγία 54 θα πρέπει να είναι κόστοβαροι να αντικατοπτρίζουν δηλαδή το κόστος παραγωγής ενέργειας, να αποκλείουν σταυροειδείς επιδοτήσεις για να δημιουργήσουν δυνατότητα ανταγωνισμού. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως, επειδή ταυτοχρόνω στα τιμολόγια είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, για να δημιουργήσουμε συνειδήσεις στους καταναλωτές προς αυτήν την κατεύθυνση με ποιο τρόπο και αν σκοπεύετε να εξετάσετε τη δημιουργία μιας συνέργειας ανάμεσα στην προώθηση των στόχων της ενεργειακής ε, αποδοτικότητας και τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας με ναι. συγκεκριμένα κίνητρα προς τους καταναλωτές που θα μπορούν να ε, αντικατοπτρίζονται στα τιμολόγια. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο. Θα χρησιμοποιήσω την εκκληκή γλώσσα. Είναι σαφές κύριε Επίτροπε ότι δεδομένων των συνθήκων της ευρωπαϊκής οικονομίας αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να χρηματοδοτήσουμε όλη την υποδομή. όλα τα δίκτυα υποδομών για την ενέργεια είναι σε κατάσταση αναμονής και φυσικά αυτά τα οποία απαιτούνται ε, δεν υπάρχουν. Αν δούμε τα αριθμητικά στοιχεία, ε, έχουμε μία εκτίμηση 400 εκατομμυρίων ευρώ, 200 εκατομμύρια ευρώ για την ε, αποθήκευση, και μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι στόχοι της των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από σήμερα μέχρι το 2020. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν ε, την όθηση για καλύτερα επενδυτικά προγράμματα για να έχουμε την υποστήριξη που, που πρέπει. Μπορούμε να σκεφτούμε με διάφορους τρόπους. ε, ε ιδιωτικέ επενδύσεις, συνταξιοδοτικά ταμεία, ε, επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Γνωρίζουμε από τις πληροφορίες που διαθέτουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου το ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει στοιχεία για να δει πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ε, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Η ερώτηση μου είναι εξή. Εμείς θα μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε ως Κοινοβούλιο επ' αυτού ή απλώς ε, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου. Άλλους 12 ομιλητές έχω. Ένα λεπτό παρακαλώ ο καθένας για να προλάβουμε. Κύριε Κωστέτ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ πολύ σύντομη. Κύριε Επίτροπε, επιμένουμε πολύ στην ενεργειακή αποδοτικότητα και βλέπουμε ότι είναι πιο δύσκολο να επιτύχουμε το στόχο που έχει καθοριστεί. Μήπως πρέπει να συζητηθεί εκ νέου αυτός ο στόχος, να προτείνουμε καινοτόμε λύσεις όπως η ε, εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τους στόχους μας. Μήπως πρέπει να προωθήσουμε τις επενδύσεις στις υποδομές βασιζόμενες σε τομεακούς στόχους Παραδείγματο χάρη υπάρχει τεράστιο δυναμικό για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει μόνο με δημόσια χρηματοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη την θέση σας επ' αυτού. Και κλείνοντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι ο ρόλος σας στο πλαίσιο της ενεργειακής στρατηγικής μέσα στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Ευχαριστώ. Ε, Ματίας. Κυρία Ματίας, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση σας εδώ. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα το οποίο έθιξε η κυρία Γκροστέτ. Έχουμε όλη αυτή τη συζήτηση για την ενεργειακή αποδοτικότητα πρόκειται για μια προτεραιότητα μόνιμη ή τουλάχιστον έτσι μας παρουσιάζεται συνεχώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, υπάρχουν ανισότητες μεταξύ ε, των δηλώσεων που αφορούν το στόχο και ε, την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής αποδοτικότητας και αυτού που γίνεται στην πραγματικότητα. Άκουσα τον Επίτροπο να λέει ότι συμφωνεί απολύτως με την Ουγγρική Προεδρία ως προς το γεγονός ότι πρέπει να ε, έχουμε μια πιο ευρωπαϊκή πολιτική για το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Εγώ θα σας αντιστρέψω αυτό το αίτημα υποστήριξης ε, και θα σας πω κατά πόσον μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο περαιτέρω, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θελοντικό καθεστώς το οποίο δεν επαρκεί. Έχουμε υποσχεθεί ένα στόχο του 20% μέχρι το 2020 για την ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά διαπιστώνουμε ότι ε, πόρο απέχουμε από αυτόν τον στόχο. Επομένως το θέμα εξακολουθεί να είναι σε κρεμότητα και δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές όπως θα θέλαμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα... Έχω μία ερώτηση για την αποδοτικότητα. Κύριε Επίτροπη, πριν από αρκετές εβδομάδες μας υποσχεθήκατε ότι θα συνεργαστείτε με τις κυβερνήσεις ώστε στο Συμβούλιο ε, να έχετε στα συμπεράσματα αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων κάποια σαφή θέση για τις δημόσιες προμήθειες. Διαβάζοντας ε, την πρόταση ε, ως έχει αυτή τη στιγμή, λέει ότι οι κυβερνήσεις θα προχωρήσουν το θέμα των δημοσίων προμηθειών νέων κτηρίων. Είναι γελίο κάτι τέτοιο. Πριν από κάποιους μήνες ψηφίσαμε μια οδηγία η οποία ούτως ή άλλως τους υποχρεώνει να έχουν ενέργεια κοντά στο μηδέν. Πώς την ερμηνεύετε εσείς αυτή τη φράση. Για μένα είναι μια κενή φράση που απλώς ζητά από τις κυβερνήσεις να τηρήσουν τον νόμο. Δεν είναι ηγετικός ρόλος αυτός. Δεύτερον, να συνεχίσω από την ιδέα της κυρίας Πιλάρντε Καστίγιο Χρειαζόμαστε καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να επιτρέπουμε να επιτρέψουμε επενδύσεις και νέους φορείς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κυρίως για χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία που έχουν δυνατότητες αλλά ταυτόχρονα βιώνουν και μια κρίση. Ε, στο σχέδιο που θα παρουσιάσετε εσείς την επόμενη Δευτέρα για τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πολύ αδύναμο, δεν έχει μεγάλη ουσία. Τι ακριβώς προτείνετε, λοιπόν για να έχουμε πρόσβαση σε κεφάλαιο, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάρμς. Ευχαριστώ. Δεν είμαι συνηθισμένη στην καινούργια αυτή αίθουσα, γι' αυτό άρχισα να ανοίξω το μικρόφωνο. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Επίτροπε, που αναφέρατε ότι το Συμβούλιο θέλει να αποφασίσει και για το ΙΤΕΡ. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, που τα διάβασα πολύ προσεκτικά, ε, δεν το είδα. Σε ποιο σημείο υπάρχει αυτή η απόφαση και τι ακριβώς θα αποφασίσετε για το ΙΤΕΡ. συνάδελφος Γκλάντε. Συμφωνώ με κάποια από αυτά που ελέγχθησαν. Η επενδύσεις αυτές πώς πόσο επιβαρύνουν το περιβάλλον. Μιλάμε για τεράστιους αγωγούς, μιλάμε για τεράστιες αποστάσεις που θα συνδέσουν τα δίκτυα αυτά. Αυτά πόσο θα επιβαρύνουν τα πράγματα. Δε, και δεν ξέρω, θα έπρεπε με τα κράτη-μέλη να φτιαχτεί μια κάποια, ε, ένας κάποιος κατάλογος με ιεραρχημένες προτεραιότητες ε, με τα κράτη-μέλη να φτιαχτεί ο κατάλογος αυτός. Και κάτι τι άλλο έχουν γίνει συζητήσεις για το τι θα γίνει με τα τέλη που επιβάλλονται για κάποια δίκτυα και δεδομένου ότι τα δίκτυα αυτά είναι διασύνοριακά, ε, δεν είναι μόνο εθνικά. Αγγέλικα Νίμπλε, θέλω να ρωτήσω κάτι κύριε Επίτροπε. Ε, είπατε ότι στις 4 Φεβρουαρίου θα πρέπει να δοθεί κάποιο πράσινο φως για εξευρωβαϊσμό από τα κράτη-μέλη. Ε, ωραία, αυτό είναι μια γενική αρχή. Πιο συγκεκριμένα πώς θα γίνει αυτό. Η κυρία Τζαβέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπο, ευχαριστούμε που είστε ξανά μαζί μας <clears throat> και θα ήθελα να σας συγχαρώ πραγματικά για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει. Δεν είναι φιλοφρόνηση. Δούλευα 15 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα στην ενέργεια και μπορώ να εκτιμήσω τη δουλειά ενός επιτρόπου. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Ε, τα ερωτήματα που θα ήθελα να σας θέσω είναι τα εξής. Ε, κυρίαρχο θέμα για την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής αγοράς είναι ο προμηθευτής. Η Ρωσία είναι και θα παραμείνει μέσω πρόθεσμα ο κυρίαρχος προμηθευτής μας στις εξωτερικές μας σχέσεις υπάρχει μία άμβλυνση θεαματική των σχέσεών μας με τη Ρωσία. Θα ήθελα την άποψή σας, πώς το βλέπετε αυτό, εάν πέραν ε, του one-way ε, σχέση που έχουμε με την Ρωσία ως κυρίαρχο προμηθευτή μας, έχουμε αναπτύξει και άλλες σχέσεις με τη Ρωσία, οι οποίες θα εξαρτήσουν τη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να υπάρχει ε, μια αλληλεπίδραση των δύο οικονομιών. Ε, και το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Στην έρευνα περιλαμβάνεται η εξόριξη. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις και για το shale gas και για την εξόριξη αερίου. Ευχαριστώ. Κυρία Κολάρσκα-Μπομπίνσκα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Θα ήθελα να μάθω την άποψή σας για την αλλαγή του ποσοστού της μείωσης ε, των εκπομπών από το 20% στο 30%. Η συζήτηση είναι ανοιχτή και ερίζουν οι απόψεις επί του θέματος. Και έχει σχέση με αυτό και η έναρξη του τρίτου σταδίου του ε, συστήματος ανταλλαγής εκπομπών. Η συζήτηση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε και για την αρχή του benchmarking ε, σε αυτή τη συζήτηση. Μιλάω για ένα νέο όριο για όλες τις χώρες που θα βασίζεται στο φυσικό αέριο. Τι άποψη έχετε εσείς από αυτού. Δεύτερη ερώτηση. Το πακέτο των υποδομών. Εμείς στην έκθεσή μας ε, υποστηρίξαμε ένα νέο κριτήριο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τα προγράμματά μας. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ένας νέος κατάλογος ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κάποιες επενδύσεις θα πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο Πρόκειται για τις επενδύσεις οι οποίες δεν θα πληρούν τα νέα κριτήρια. Το σχέδιο του Nord Stream ε, πληρεί τις νέες προϋποθέσεις, παραδείγματος χάρη το κριτήριο της διαφοροποίησης. Νομίζω ότι δεν το πληρεί. Επιπλέον, το, εξυγχρονισμός των παλιών ενεργειακών δικτύων. Νομίζω ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν, διότι τα νέα στοιχεία δεν μπορούν να συγχωνευτούν με κάτι παροχημένο. Ο κύριο Σόουσα Βάγνερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα για να θέσω την εξή ερώτηση στον Επίτροπο, όπω και αρκετοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε ποιο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για την ανακοίνωση για τις ε, προτεραιότητες στην ενέργεια σε θέματα χρηματοδότησης των προγραμμάτων. Νομίζω ότι επί του θέματος θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι ευπρόσδεκτη από πλευράς ευρωβουλευτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νταντζέλης, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ότιγκερ για την παρουσία του εδώ μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την ενεργειακή πολιτική. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία μιας νέας αγοράς ενέργειας είναι απαραίτητη κυρίως για να μπορέσουμε να υπερκεράσουμε τις εθνικές αγορές, ε, στις οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει μία επιχείρηση η οποία ασκεί μονοπόλιο. Το να μπορέσουμε λοιπόν να βελτιώσουμε την ε, ενεργειακή αγορά θα έχουμε σίγουρα σημαίνει ότι θα έχουμε σίγουρα μεγαλύτερε επενδύσει για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας και θα είναι καλύτερε οι συνθήκε τη αγορά για του καταναλωτέ. Μεγαλύτερη συνέργεια λοιπόν για μεγαλύτερη προστασία των τιμών, ιδίω για τι επιχειρήσει και του καταναλωτέ. Να περάσω τώρα εντάχει στις δύο μου ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το τρίτο πακέτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μπορεί να διασφαλίσει ότι η ε, απελευθέρωση που προβλέπεται θα διασφαλίσει ότι οι εθνικοί ρυθμιστές θα εργάζονται κατά τρόπον ώστε να έχουμε ασφάλεια στην ενέργεια και αποδοτικότητα της ενέργειας. Ε, δεύτερον, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών ε, κατά 20% μέχρι το 2020. Πώς σκοπεύετε να διευκρινίσετε τους τρόπους χρηματοδότησης των τεχνολογιών που θα μας επιτρέψουν να επιτέχουμε τη στρατηγική του 2020. Κυρία Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σαφώς θα είναι πολύ σημαντικό το Συμβούλιο αυτό, κύριε Επίτροπε. Γι' αυτό και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για το γεγονός ότι μας διαβιβάσετε τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία θα συζητηθούν, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Δύο ερωτήσεις για σας. Η πρώτη αφορά το θέμα της έρευνας και της καινοτομίας. Σαφώς οι περισσότερες ε, ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι και τα θέματα που θίξατε εσείς ε, σημαίνει ότι θα έχουμε τεχνολογικές ε, προόδους και καινοτομία. Αναφέρατε ότι θα συζητηθεί και σε αυτό το Συμβούλιο το θέμα, Βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία όπου καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για το νέο πρόγραμμα πλαίσιο, το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, οι οποίες θα έρθουν επισήμως στο Κοινοβούλιο σε ένα-δυο μήνες. Θα μπορούσατε να μας πείτε ένα-δυο πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, τι ακριβώς θα θεωρήσετε προτεραιότητα, θα πρέπει να βελτιωθούν οι επενδύσεις, ε, ε πώς θα το συντονίσετε με την Επίτροπο Γκέν και Επίσης, ένα άλλο θέμα. Ε, ξέρετε ότι λόγω καταγωγής ε, και επειδή ακριβώς θέλουμε μία ε, πιο αποδοτική αγορά ενέργειας, με ενδιαφέρει το θέμα των υποδομών. Και νομίζω ότι θα ενδιαφέρει και τους συναδέλφους να ακούσουμε κάτι παραπάνω επί του θέματος. Πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε το θέμα και τι αποτελέσματα περιμένετε από τις διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι εξελίξει αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ, Επίτροπε. Θέλετε να επιταχύνετε την εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς, το τρίτο πακέτο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερες διαδικασίες επί παραβάση κατά των κρατών μελών ή περισσότερη νομοθεσία. Για τις υποδομές, σωστά υπογραμμίζεται πόσο σημαντικές είναι οι επενδύσεις. Όμως, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόσκομα για τις επενδύσεις και τις υποδομές μας, το γεγονός ότι δεν έχουμε συνένεση για το ε, σχεδιασμό ή είναι η χρηματοδότηση το πιο σοβαρό πρόβλημα. Αναφερθήκατε επίση στην έρευνα για την ενέργεια και υποστήριξη από τα κράτη-μέλη για κάποια προγράμματα. Συμπεριλαμβάνεται και το ίτερ, ε, θα έχει περισσότερη υποστήριξη το ίτερ. Και επειδή έχω και λίγο χρώμα ακόμα, να σας πω ότι το Ενεργειακό Φόρουμ Ενέργειας ε, ε περιμένει εναγωνίως να σας δει και στο μέλλον, στους κόλπους του. Η κυρία Καρβάγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την, τον Επίτροπο. Εχθές το βράδυ ο Πρόεδρος Ομπάμα έδωσε μια ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης και αναφέρθηκε και στις ενεργειακές πτυχές και την πολιτική ενέργεια. λέγοντας ότι η χώρα η οποία θα κατευθύνει τις πολιτικές, ε, της ενέργειας με καθαρή ενέργεια θα είναι και ο παγκόσμιος ηγέτης επί του θέματος της ενέργειας και κατά την άποψή του η χώρα αυτή θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Κατά την άποψή σας, τα συμπεράσματα του επόμενου Συμβουλίου θα μπορέσουν να χρησιμεύσουν ώστε να αυξηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ε, σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Κυρία Χούμπνερ. Χούμπνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτρόπε, ήσασταν ιδιαίτερα δραστήριο όσον αφορά την δημιουργία του Ναμπούκο και άλλων αγωγών το νότο της Ευρώπης. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τον αγωγό North Stream. Είναι ένας αγωγός ε, που περνάει από την Βαλτική και τα μεγαλύτερα σκάφη δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν ε, λιμένες στο νότο της Βαλτικής. Ένα τεράστιο πρόβλημα για την Πολωνία και τη Λιθουανία. Πώς θα προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα αυτό. Κάνετε διαπραγματεύσει για το θέμα αυτό και Πώς προτείνετε να επιληθεί αυτό το αδιέξοδο. Και μια δεύτερη ερώτηση. Έχει γίνει μια πρόταση για αύξηση κατά 100% της βιομάζας ε, στο μείγμα ε, ενεργειών. Ποια είναι η γνώμη σας από αυτού. Προσπαθούμε να βρούμε κονδύλια για την ανάπτυξη των δασών στον Αμαζόνιο, παραδείγματο χάρη. Δεν νομίζετε ότι θα είναι υπερβολικά μεγάλη η συμμετοχή τη βιομάζα στο ενεργειακό μείγμα και θα μπορούσε να δημιουργήσει ε, αποψήλωση των δασών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο να προσπαθήσει να απαντήσει. Ξέρω ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχετε στη διάθεσή σας, θα σας είμαστε ευγνώμονες όμω αν τα καταφέρετε. Der Europäische Rat το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν μπορεί να ασχοληθεί με πολλά θέματα σε λεπτομέρεια. Σε δυόμιση ώρες δεν θα προλάβει να αντιμετωπίσει όλα τα θέματα. Και οι λεπτομέρειες δεν είναι θέμα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, αλλά των εξειδικευμένων υπουργών και ομάδων εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει τις γενικές αρχές, ε, ε, απαντώ σε κάποιες ερωτήσεις που έγιναν από αυτού. Άλλα θέματα σίγουρα θα αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια του έτους με συγκεκριμένες προτάσεις και ανακοινώσεις ε, και με νομοθετικά κείμενα που θα φτάσουν και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Ενέργειας. Και για το κλίμα και για την ε, ενεργειακή πολιτική στο μέλλον είναι υπεύθυνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για την ε, βιοενέργεια είναι και αυτό ένα θέμα και εδώ έχουμε τον οδικό χάρτη για το 2050. Είναι μια πολιτική λοιπόν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για όλους τους τομείς θα έχει επιπτώσεις για την πολιτική μεταφορών, για την ενέργεια, για τη γεωργία, για τη βιομηχανία και για την αποδοτικότητα και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τη συμμετοχή των μορφών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Θα συζητήσουμε και τις θετικές εμπειρίες και τα προβλήματα και τις προτάσεις που θα αναφερθούν στα συμπεράσματα. Μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα, μας ενδιαφέρει η φόρος ανάπτυξη, ασφάλεια των ειδών διατροφής, και διατήρηση του τοπίου, γιατί δεν θέλουμε ε, να καταστραφεί το τοπίο στις ε, χώρες μας. Αυτό είναι θετικό και για τον τουρισμό, αλλά και για την ε, βιωσιμότητα των πολιτικών μας. Το θέμα του αγωγού North Stream. Νομίζω ότι θα τηρηθούν όλες ε, οι απαραίτητες διατάξεις προς όφελος ε, και της προστασίας της φύσης και του ζωικού βασιλείου και των αλλιευτικών πόρων αλλά και το θέμα της ε, πλευσιμότητας των λιμένων. Όλα αυτά θα εξεταστούν προσεκτικά μέσα στον προγραμματισμό που γίνεται και θα συνεχίσει ε, η εξέλιξη των μέτρων για τον North Stream, λαμβάνοντας υπόψη όλες ε, τις απαιτήσεις για τα θέματα αυτά. Δεν έχει πάρει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια North Stream, γιατί δεν είναι ένα πρόγραμμα σε υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λετωνία, Λιθουανία και Εστονία και η Πολωνία έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη σύνδεση με την Ευρώπη, γιατί το φυσικό αέριο από την Σιβηρία θα είναι φυσικό αέριο που θα φτάνει, για όλη την, θα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας ενδιαφέρει να συνεισφέρουμε στην διαφοροποίηση, ούτως ώστε να έχουμε πολλαπλές ε, πηγές ε, ενεργειακού εφοδιασμού και ενεργειακή ασφάλεια. Για τους ε, διαδρόμους ε, και για την, ε, τον ενεργειακό εφοδιασμό ήθελα να πω ότι προετοιμάσαμε πια ένα έτος την επίσκεψη στο Αζερβαϊτζάν με τον πρόεδρο Μπαρόζο. Χρειάζεται ένας συνομιλητής και μία υπογραφή για να μπορέσουν να γίνουν διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Μοχαντοφ, ο κύριος Σαλίεβιτς δεν ε, θα ε, βάλει την υπογραφή του κ. Καρίμοφ. Υπογράφουμε σε εγγυημένη τιμή για 30 χρόνια με μία υπογραφή. Ε, δεν είναι απόλυτα γνωστό το πώς γίνονται αυτές ε, οι αγορές. Υπάρχουν ε, πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των ε, κρατών μελών και των φορέων χρηματοδότησης και των επιχειρήσεων και είναι καθήκον μας να τα εξηγήσουμε όλα αυτά και ελπίζω ότι θα επιτύχουμε και είμαι αισιόδοξο για τη χρηματοδότηση για τα, 10, για τα δισεκατομμύρια και για τον όγκο που θα ε, εξασφαλίσουμε. Ε, έχουμε μια νέα οδό και μια νέα πηγή. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε διπλή διαφοροποίηση και ασφάλεια εφοδιασμού. Δεν μιλάω εξάλλου για τον Αμπούκο, μιλάω για τον Αμπούκο συν. Δεν μιλάμε για τον αγωγό από την ε, Βιέννη μέχρι τα σύνορα της Τουρκίας-Γεωργίας. Ε, πρέπει να έχουμε νέα κατασκευή μέχρι τον Πακού. Αγωγός μέσω της Κασπίας προς τις πηγές στο Τουρκμενιστάν και αγωγός ε, μέσω της Κασπίας θάλασσας. Πράγμα το οποίο θα χρειαστεί και αντίστοιχη υποστήριξη από πλευράς ναυσιπλοείας. και το Ιράν ε, θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Το ε, ε, Ιράκ μέσω της Βαγδάτης ούτω ώστε να έχουμε την απάντηση που θέλουμε για τον αγωγό. Ένας αγωγός θα περνάει από την Τουρκία 6 ε, σε δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσω της Τουρκίας και μέχρι την ε, Βιέννη και με ένα κλάδο προς την Ιταλία και θα ε, τροφοδοτεί και την Ιταλική αγορά και την Κεντρική Ευρωπαϊκή αγορά. Και αν δείτε ότι είναι η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία σε αυτό το σημείο πάλι εξασφαλίζουμε τον εφοδιασμό και προς αυτές τις χώρες. Και την επόμενη εβδομάδα ο κύριος Μπαρός έχει καλέσει τα κράτη Βίζεγκρατ και θα σας πω γιατί. Γιατί αν έρθει ο Ναμπούκο θα έχουμε ένα τεράστιο πλεονέκτημα ε, να έχουμε παράλληλα και τη σύνδεση βορρά-νότου. Και το φυσικό αέριο από τον αγωγό αυτό, τον Ναμπούκο Συν, ε, για την Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες θα είναι ένα πλεονέκτημα και για την ε, Κροατία και τα Δυτικά Βαλκάνια θα είναι κάτι το εφικτό. Οπότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματική ευρωπαϊκή λύση από την οποία όλοι θα μπορούν να υποφεληθούν. Άκουσα την ομιλία του Πρόεδρου Ομπάμα με δύο μικρές αντιρρήσεις για αυτά που είπε. Δεν άκουσα τη λέξη Ευρώπη πουθενά. Ε, μας θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα. Η ομιλία αυτή είναι σημαντική για το Κογκρέσο. Ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον, κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Κογκρέσο, όπως και το διοξίδιο του άνθρακος ένα θέμα που ε, τους ενδιαφέρει πολύ μετά τις εκλογές. Το σχέδιο ζήτα το συνεχίζουμε και ε, ε, στη συνεδρία της 4 Φεβρουαρίου θα παίξει σημαντικό ρόλο και η ενέργεια και η καινοτομία. Είμαστε σε επαφή και θα συνεχίσουμε με το επόμενο πρόγραμμα ε, για την ενέργεια και την έρευνα και είναι πρόθυμοι και οι αρμόδιοι για την ενέργεια και ο πρόεδρος Μπαρόζο επίσης και θα δοθεί ε, αυξημένη χρηματοδοτική σημασία μέσα στην Επιτροπή. Είναι κάτι για το οποίο αγωνίζομαι. θα χρησιμοποιήσει το ίτερ όλα τα διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης και θα αποφασιστεί το πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση και θα είναι θέμα του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να κάνουμε διαπραγματεύσεις ε, και με το Πεκίνο και με την Ουάσιγκτον για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις προτεραιότητές μας. Η Κομισιό ε, και η Γαλλία μπορεί να είναι υπεύθυνη ε, για τις διαπραγματεύσεις. Και το ίτερ δεν είναι μόνο ενεργειακά προγράμματα. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συνολικά, μια εταιρική σχέση. Και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Το θέμα συζητείται με δημοκρατικές διαδικασίες και από την πλειοψηφία. Εγώ το είτε το βρήκα. Υπήρχε ήδη και δεν θέλουμε να το εγκαταλείψουμε. Δεν θέλουμε το ίτερ να καταναλώσει αυτά τα οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει και κάτι άλλο. Και προσπαθούμε προς όλες τις κατευθύνσεις να κινηθούμε. Τώρα για τα κριτήρια των υποδομών, τις προτεραιότητες, θα τις θέσουμε ως δεύτερο βήμα το καλοκαίρι. Η Ευρώπη ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά. Μιλάμε για την ε, συμμετοχή, στη συνέχεια έχουμε την αξιολόγηση αυτών που γίνονται και μετά περνάμε στο επόμενο βήμα και θα φτάσουμε το καλοκαίρι σε αυτό το επόμενο βήμα με συγκεκριμένε προτάσεις για τη χρηματοδότηση και με το κατάλογο προτεραιοτήτων. Και θα ξαναείμαι εδώ να τα ξανασυζητήσουμε. Πολύ σωστά μιλάτε για καινοτόμες προτάσεις ε, χρηματοδότησης δεν έχουμε κανένα μηχάνημα που να παράγει χρήματα. Πρέπει να βρούμε λύσεις εφικτές ως προς τη χρηματοδότησή τους. Πρέπει να είμαστε καινοτόμοι και να μας εμπιστεύονται και οι αγορές. Μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά δεν είναι φιλανθρωπική οργάνωση. Ε, πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ορίσουν το πόσο θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη χρηματοδότησή της. Και θα είναι τέρος μας για τα προγράμματα υποδομών η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία προτείνει η Επιτροπή και από τα μέσα ενημέρωσης και από τις χώρες. Και η Γερμανία ξέρω ήταν επικριτική σε αυτά τα οποία ε, συζητήθηκαν. Υπάρχουν τα τρέχοντα καθήκοντά μας και παράλληλα με αυτά θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και επιπλέον ζητήματα υποδομών. Πάντως η ενέργεια είναι σε σημαντική προτεραιότητα η ενέργεια ε, και οι μεταφορές και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι τρεις τομείς υποδομών ε, στους οποίους ε, αναζητούμε καινοτόμα εργαλεία και ιδιωτικό κεφάλαιο. Και αν συμμετέχουν και συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλοι χρηματοδοτικοί φορείς, ο σκοπός είναι να μην είναι κάτι το οποίο θα είναι περισσότερο δαπανηρό ένα ασφαλιστικό ταμείο, ένα συνταξιδοτικό φορέας ε, θα θέλει να έχει υψηλότερου ε, τόκους από ό,τι θα έβρισκε στην ε, αγορά κεφαλαίων. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να τους προσφέρουμε αξιοπιστία για να επιλέξουν εμά για επενδύσει. Και τίθεται το ερώτημα του τι χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό και τι από τον δημόσιο τομέα και στο ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο θα πρέπει να θέλουν να επενδύσουν οι ιδιοκτήτες ε, δικτύων ε, και να θέλουν να το πληρώσουν οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές θα το πληρώσουν τους ή άλλως, είτε διότι χρησιμοποιούν το ρεύμα, γιατί ε, όλοι ε, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το τομέα του, του ηλεκτρισμού πληρώνουν για τη χρήση του, του, ηλεκτρισμού. Μιλάμε για ε, δίκτυα από τη μια άκρη στην άλλη από τη μια άκρη της Ευρώπης στην άλλη. Υπάρχουν όμως ε, ε, ε, δίκτυα που δεν είναι τόσο αποδοτικά. Και ξέρουμε ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορεί σε, κάποιο, σε κάποια γραμμή να είναι και επιζήμιες. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε προγράμματα συγχρηματοδότησης και μιλάμε για προγράμματα τριετή με 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τις διασυνδέσεις. Και θα χρειαστούν 5 έως 10 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση όλων των σημαντικών αγορών η ολοκλήρωση των ε, επιμέρους αγορών μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το 2050. Δεν μπορεί καμία χώρα μόνη της με την αγορά ηλεκτρισμού και ε, φυσικού αερίου να μείνει έξω από την ε, ευρωπαϊκή αγορά. Και ελπίζουμε ότι μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια θα καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς. Πιστεύω ότι είναι πολύ υψηλή η πιθανότητα επιτυχίας αυτών τα οποία ε, ε, τώρα ε, προτείνουμε. Και για το διοξίδιο του άνθρακου θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν τέλη και φόροι και υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορούμε να προτείνουμε και ίδιους πόρους για να μην υπάρξουν ε, καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο χωρίς να υπάρχει ε, όφελος ε, για το περιβάλλον και για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε το δεύτερο και το τρίτο ενεργειακό πακέτο, πριν περάσουμε σε τέταρτο ενεργειακό πακέτο. Να ολοκληρώσουμε το δεύτερο και να περιμένουμε και από τα κράτη-μέλη το τι θα κάνουν για το τρίτο με διαπραγματεύσεις και με συνέχιση των συζητήσεων. διαπιστώνουμε και στα κράτη-μέλη ότι μια σταθερή τιμή για το ρεύμα ή για το φυσικό αέριο ή μια μειούμενη τιμή είναι πολλές φορές ε, τμήμα ε, της ε, πολιτικής είτε της οικιστικής πολιτικής είτε των μέτρων που προτείνουν οι κυβερνήσεις στους πολίτες τους. Χρειαζόμαστε διαφάνεια και πλήρη κάλυψη του κόστους για την ενεργειακή αποδοτικότητα θέλουμε καταρχήν να υπάρχουν ξεκάθαρες προτάσεις, ξεκάθαρα σχέδια. Και στις 2 Μαρτίου θα υποβάλουμε την πρότασή μας και το Μάιο θα κάνουμε και μια περαιτέρω συζήτηση για τα επόμενα βήματα. Για τις σημαντικές επενδύσεις, για τα υπάρχοντα κτίρια, προσπαθούμε να έχουμε άνοιγμα των περιφερειακών προγραμμάτων προς αυτήν την κατεύθυνση. θέλουμε να προχωρήσουμε με την ανακαίνιση ε, και την εξυγίανση των υπαρχόντων κτηρίων πριν περάσουμε σε άλλα σχέδια και χρηματοδοτούμενα προγράμματα για μαρίνες ή για οτιδήποτε άλλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. την επόμενη Δευτέρα θα υποβάλουμε μια νέα πρόταση, Τόμας, και νομίζω ότι θα έχετε την ε, ευκαιρία ε, να την ε, ακούσετε προς τον κύριο Τούρμες. Θα έχουμε πολλές δομές χρηματοδότησης, οι οποίες μπορούν να... Μπορεί να τη δείτε μέσα στην ανακοίνωση και από εκεί πέρα μπορούμε να τη συζητήσουμε. Μιλάμε ε, για προγράμματα ε, για αεολικά πάρκα offshore και ε, για ολοκλήρωση αγορών Ολλανδίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας για να δούμε πού μπορούν να γίνουν οι επενδύσεις και μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι υποδομές που μπορούν να συντονιστούν ε, ανάμεσα στις διάφορες χώρες, ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία παραδείγματος χάρη. Και οι Ευρωπαίοι Ευρωβουλευτές είναι οι καλύτεροι Ευρωπαίοι που μπορούν να προωθήσουν το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεν ε, θα προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα, θα προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές λύσεις και στην ε, Τινησία, αν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση ε, στην ε, Τινησία ή δημοκρατικές κυβερνήσεις στην Βόρεια Αφρική, στις χώρες του Μαγκρέμπ, μας ενδιαφέρει να έχουμε εταιρική σχέση μαζί τους και εταιρική σχέση μαζί τους και στον τομέα της ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε και για να το έχουμε αυτό θα χρειαστούμε επενδυτές, ε, ευρωπαϊκά δίκτυα και θα χρειαστούμε ε, και προτεραιότητα ε, σε ευρωπαϊκές λύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θα προωθήσουμε τις ε, εφικτές ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, σε λογικές τιμές. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες σας τις ερωτήσεις και θα έχουμε και περισσότερες ευκαιρίες να συζητήσουμε λεπτομερέστερα θέματα. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις εξαντλητικές σας απαντήσεις. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω που ήρθατε να μας επισκεφθείτε πριν από το Συμβουλίο των Υπουργών. Είναι καινούριο αυτό να έρχεται ο, Υπουργό, ο Επίτροπος εδώ πριν να πάει στο Συμβούλιο των Υπουργών για να μας παρουσιάσει το τι θα γίνει στο Συμβούλιο και να μπορούμε να το σκεφτούμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Οιτιγκέρ. Ωραία λοιπόν. Προχωρούμε ε, ολοταχώς στα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης ε, τα οποία θα πρέπει να τα διεκπαιρεώσουμε πάρα πολύ γρήγορα διότι έχει ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε στο τέος 9 μην 6, 6 τη διάταξη. Ο Ευρώπη ο πρώτο τουριστικό προορισμό Η συγγητή είναι ο κύριος Χατζημαρκάκης. Να είμαστε σύντομοι. Ένα λεπτό περιμένετε να φύγουν αυτοί που φεύγουν από την αίθουσα να επικρατήσει μια κάποια ησυχία. Meine Κυρίες και κύριοι, δεν μπορείτε να βγείτε γρήγορα από την αίθουσα να κάνετε ήσυχια για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα επόμενα θέματα της σημερινής διάταξης. Συγγνώμη, ναι, αλλά βιαζόμαστε. Άμα θέλετε να φύγετε, φύγετε, αλλά όχι. Αλλά με ησυχία όμως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα πράγματα θα πάνε σχετικά γρήγορα. Το θέμα είναι αν θέλουμε να αναπτύξουμε την Ευρώπη ως τουριστικό προορισμό ή όχι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρώτη συζήτηση που έγινε ήδη εδώ στην Επιτροπή στις αρχές του Δεκέμβρη. Ευχαριστώ λοιπόν α, για αυτά που ελέγχθησαν εκεί και για τις προτάσεις που έκαναν οι συνάδελφοι. Τις περισσότερες προτάσεις τις ενέταξα στο κείμενο. Δεν έχω πολλά πράγματα να συμπληρώσω. Λέω βεβαίω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει επιπλέον αρμοδιότητες στον τουρισμό και ο Επίτροπος Ταγιάννη έχει αναλάβει τις σχετικές αρμοδιότητες και θέλει να υποστηρίξει την Ευρώπη σαν πρώτο τουριστικό Προορισμό. Σημαντικό ρόλο παίζει εδώ η εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε προσωπικό εκπαιδευμένο με ψηλά, ψηλό επίπεδο προσόντα για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τουρίστες και από το ιστορικό της Ευρώπης αλλά και εκτός Ευρώπης. Τα standards πέρσι αλλάξανε δηλαδή και χρειάζεται εδώ να δούμε και την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων στον τομέα των τουριστικών σπουδών. Εν τω μεταξύ ε, υπάρχουν πολλά ε, ιδιωτικά προγράμματα ανταλλαγών που ε, λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη και που είναι πάρα πολύ επιτυχή. Πάρα πολύ νέοι και από την Ευρώπη και ε, αλλά και εκτός Ευρώπης έρχονται στην Ευρώπη και κάνουν ανταλλαγές με τους Ευρωπαίους. Πολύ καλά προγράμματα ανταλλαγών λοιπόν. Επίσης, ε, άμα θέλουμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό θα μπορούσαμε να φανταστούμε ε, ένα ενιαίο είδος μάρκετινγκ στην Ευρώπη μέσω του διαδικτύου δεν ξέρω αν θυμάστε παλιότερες διαφημίσεις από την Ιαπωνία ή από την Κίνα και ε, όπου εκεί προ διαφημιζόταν ας πούμε μεγάλες ομάδες Ασιατών οι οποίοι ερχόταν στην Ευρώπη και βλέπανε την Ευρώπη σε μια εβδομάδα. Αυτό προϋποθέτει ένα κοινό ο, marketing το, και κοινέ διαφημίσεις οι οποίες πρέπει να προωθήσουμε όχι μόνο στην Ασία αλλά και στη Βραζιλία, Ινδία κτλ. Ε, επίσης ιατρικός προορισμός ε, τουρισμός υγείας ε, ας πούμε ε, είναι γνωστό τι όλη η Ευρώπη σαν τουριστικός προορισμός για θέματα που σχετίζεται με θέματα υγείας Μιλάω για ένα τουρισμό που σχετίζεται ή με πραγματικά θέματα υγείας και περίθαλψη νοσοκομιακή κτλ. ή με θέματα spas, wellness κτλ. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα, ένα σήμα, αν θέλετε, τουριστικό σήμα για την Ευρώπη. Ε, ένα κιανού σταυρό, κατά κάποιο τρόπο, ε, θα μπορούσαμε να φροντίσουμε να εξασφαλίζουμε υψηλά στάνταρτς, να, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε με κονδύλια από τη συνοχή ε, ε, και βεβαίως δεν θα πρέπει να δίνουμε στο τυφλά κονδύλια, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε και να ε, διαβεβαιώνουμε ότι τηρούνται κάποια standards. Από εκεί και πέρα, στο τομέα της απασχόλησης θα πρέπει να δούμε το νομοθετικό πλαίσιο των ε, όρων εργασίας. Ε, γιατί εδώ στον τουρισμό έχουμε πολλές υπερορίες, έχουμε δουλειά τη Σαββατοκύριακα και Ε, και δεν πρέπει να τα ξεχνούμε αυτά. Τελευταίο θέμα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ή να εγγυόμεθα αν θέλετε την, ή να βελτιώσουμε την ασφάλεια των ταξιδιωτών, των τουριστών που έρχονται εδώ στην Ευρώπη. Ε, δεν είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, αλλά επειδή υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα, νομίζω ότι αν προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μια νεοποίηση, ομογενοποίηση κατά κάποιο τρόπο, αυτό θα μας βοηθήσει. Ο κύριος Μεζάρος. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ και τον κύριο Χατζημαρκάκη για την παρουσίασή του. Όντως το θέμα του τουρισμού μας ενδιαφέρει και βεβαίως ξέρουμε ότι ο Ανάπτυξη Ευρώπης ως τουριστικό προορισμό θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας αλλά γι' αυτό πρέπει να εξυγχρονίσουμε και τις υπηρεσίες μας να προωθήσουμε τον τουρισμό μας. Ξεκίνησαν όλα αυτά από το 2008 ε, για την προσέλκυση νέων τουριστών εδώ στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι ήδη η Ευρώπη είναι ένα σημαντικός τουριστικός προορισμός. 1,8 ε, εκατομμύρια μισοδήματα πλήρους απασχόλησης ε, ισοδύναμα πλήρως απασχόληση εργάζονται για τον τουρισμό στην Ευρώπη υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό με άλλα λόγια που θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και θα πρέπει να τονίσουμε ορισμένα α, θετικά, ορισμένες ιδιαιτερότητες που έχει η Ευρώπη. Αναφέρθηκε ο κ. Χατζημαρκάκης στον α, α, τουρισμό σε σχέση με την υγεία είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομ, συγχρόνως μπορούμε να προωθήσουμε και άλλες πτυχές της, Ευρω... της Υπήρου μας, της παραδόσεις μας, της χριστιανικές μας ρίζες και τα λοιπά για να προσελκύσουμε ε, περισσότερους τουρίστες οι οποίοι να περάσουν καλά στις χώρες μας. Πράγματι χρειάζεται ένα ε, κοινό μάρκετινγκ και ένα κοινό σήμα για την Ευρώπη. Βεβαίως και βεβαίως θα πρέπει να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε οποιασδήποτε κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να προωθηθεί ο τουρισμός. Ευχαριστώ κύριε Φρανκό. Ω σκιώδη ηγητή για το ΕΛΚ, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση που αποτελεί πολύ καλή βάση εργασία και συζήτηση. Ο τουρισμό είναι ένα παράγον δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει οι χώρε μα να προσαρμοστούν σε νέε τουριστικέ ροέ που προέρχονται από τι αναδυόμενε χώρε που βρίσκονται σε οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα με την τεχνολογική ανάπτυξη και με τη χρήση της πληροφορικής και του διαδικτύου και με προστασία του περιβάλλοντος δημιουργούνται νέες ανάγκες και τα επαγγέλματα του τουρισμού θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες ανάγκες. Νέε τουριστικές προσφορές, εναρμονισμένες με τη φύση περισσότερο από ό,τι πριν, προωθώντας τι ε, αξίες ε, της υπαίθρου σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να αποκτήσουν προτεραιότητα και θέλουμε να προωθήσουμε μορφές όπως τουρισμός στο αγρόκτημα ή τουρισμός σε μικρά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή τουρισμός υγείας ε, με βάση τις δημογραφικές εξελίξεις. Αυτές είναι οι νέες μορφές σύγχρονου τουρισμού που πρέπει να τις ενθαρρύνουμε για να προωθήσουμε ένα τουρισμό που θα σέβεται την πολιτισμική μας πολυμορφία και τις ιδιαιτερότητες των πολιτών μας έχω διάφορες προτάσεις. Να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό και μεσογειακό παρατηρητήριο τουρισμού που θα καταγράφει τις επιδόσεις του τομέα και θα ασχολείται ιδιαίτερα με την ανταλλαγή καλών πρακτικών για τις νέες μορφές βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού. Ακόμη θα πρέπει στο μελλοντικό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και ε, καινοτομίας να μπει μια σημαντική πτυχή τουρισμού και θα πρέπει να τονίζουμε τις νέες τεχνολογίες, ιδίως αυτές που δημιουργούν εξοικονόμηση ενέργειας και που είναι θετικές για το περιβάλλον πειραματισμό με νέε μορφές βιώσιμου τουρισμού σε συγκεκριμένε γεωγραφικέ ζώνες για να μπορέσουμε ε, να εξισορροπήσουμε τον τουρισμό που είναι πολύ επικεντρωμένο στι παράκτιε ζώνες θα δώσουμε σημασία και στις επιπτώσεις ε, του τουρισμού και θα δουλέψουμε πάνω στον ε, τουρισμό προσπαθώντας να σπάσουμε την εποχικότητά του ε, και θα επιμείνουμε στην κατάρτιση και γλωσσική κατάρτιση και χρήση του διαδικτύου καθώς και θα προσφέρουμε εξειδικευμένα μεταπτυχιακά διπλώματα για τον τουρισμό όπως το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο ακόμη θα χρηματοδοτήσουμε πειραματισμού σε, νέες, σε νέους προορισμούς. Αυτά θα οδηγήσουν σε καλύτερη ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού κλάδου. Ακόμη θα προτείνω μία τροπολογία για την πρόθεση του επιχειρηματικού και του συνεδριακού τουρισμού, για την ένας τομέας με πολλές θετικέ επιπτώσεις για τις ε, κοινότητες σε τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη. Επίσης, επιμένουμε στην ελκυστικότητα των ε, υπερπόντιων διαμερισμάτων, γιατί ε, είναι μία εναλλακτική λύση και για τους πολίτες των ΗΠΑ και για πολίτες χωρών όπως η Βραζιλία, που έχουν ανερχόμενο εισόδημα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρέιρα Μαντουρέλ, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του και να του τον ευχαριστήσω διότι στην πρόταση έκθεσής του συμπεριλάβε και κάποιες από τις προτάσεις μας ε, και έκανε μια καλή ανταλλαγή απόψεων μαζί μας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες σκέψεις. Θα ακολουθήσω την ε, σειρά που έχει ακολουθήσει και ο εισηγητής ε, στην εκθεσή του. Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται στην ε, ανταγωνιστικότητα του της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να κάνουμε σαφή σύνδεση της ανταγωνιστικότητας με το να ενδυναμώσουν ε, την, ε, ε, τις επενδύσεις γιατί θέλουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί και με καινοτόμα μέσα και όχι μόνο μειώνοντας τις τιμές. Το θέμα της καινοτομίας δεν προκύπτει πουθενά στην έκθεση. Ως Επιτροπή Ήτρου Ήτρε, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, να λέμε συνεχώς ότι πρέπει να δώσουμε δυνατότητες να υπάρχουν καινοτομίες ε, ε, και κυρίως στον ευρωπαϊκό τουριστικό τομέα, διότι μας δίνει πολύ καλά αποτελέσματα για ένα κλάδο ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για το ΑΕΠ μας. Και επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε να θεμελιώνουμε την ε, καινοτομία στην Ευρώπη. Το αναφέρει ο εισηγητής, αλλά δεν υπάρχει κάπου ρητή αναφορά στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας για τον ε, τομέα αυτό. Ιδίως ε, επειδή θέλουμε να έχουμε τη βέλτιστη δυνατή προσαρμογή της προσφοράς στις νέες ανάγκες για να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικασίες και να έχουμε καλύτερα προϊόντα προς όφελος των καταναλωτών. Όσον αφορά τώρα τη βιωσιμότητα του κλάδου, ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 2 από τον εισηγητή, θεωρώ ότι είναι απαραίτητη ε, ως ένα καλύτερος συντονισμός, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσουμε νέες δυνατότητες για μεταφορά τεχνολογίας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε νέα μέσα και να καινοτομήσουμε προκειμένου ο τομέας να βελτιωθεί σε στρατηγικού τομείς όπως είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Και τέλος, ε, θεωρώ ότι θα άξιζε τον κόπο να τονίσουμε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο, ο, ο τουριστικός τομέας στην βιομηχανική μας πολιτική, να τονίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου, όπως είναι η εποχικότητα για παράδειγμα, ε, ο εισηγητή ε, ανέφερε ότι έχουμε ένα ευέλικτο πλαίσιο και θα πρέπει να καινοτομήσουμε, να έχουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίε και να εμείνουμε στην ε, συνεχή επιμόρφωση. Το αναφέρει ο εισηγητή και επιμένω κι εγώ γιατί θεωρώ ότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να είμαστε ανταγωνιστικοί από πλευρά ποιότητα και θα πρέπει να αναφέρεται αυτό ρητό στην έκθεση. Θα πρέπει να πω ότι συμφωνούμε απολύτω με τι σκέψει του εισηγητή όσον αφορά το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στην, στον τουριστικό κλάδο και να πω ότι μου άρεσε και πάρα πολύ η ιδέα του συναδέλφου που ανέφερε ότι θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη γραμμή στο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομία για τον τουρισμό. Ω και όδηση ολοκληρώνοντα, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μου θα παρουσιάσει κάποιε τροπολογίε, κυρίω λαμβάνοντα υπόψη αυτά που μόλι σα ανέφερα, Τροπολογίε που είμαι βέβαιη ότι θα είναι ευπρόσδεκτε από τον εισηγητή και από τι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφος Όντι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για τις προτάσεις του. Και προτείνω να επιμείνουμε στον τουρισμό ε, που έχει σε στόχο την ευημερία και τις ε, ιαματικές πηγές. Οι ιαματικές πηγές ε, κυρίως επικεντρώνονται σε περιοχές που έχουν και αρχιτεκτονικά πλούσιο παρελθόν και νομίζω ότι μπορούμε να το προσφέρουμε ως ευρωπαϊκή μορφή τουρισμού οι Κινέζοι έχουν εγκαταλείψει αυτές τις δραστηριότητες και οι Αμερικανοί το ίδιο. Ξέρουμε ότι οι Ρωμαίοι άρχισαν να δημιουργούν τέτοια δίκτυα θερμών ε, πηγών και έχουμε και σχετική πρόταση και για τους φίλους τους Ουγγρους με τον πλούτο τέτοιων πηγών που έχουν στη Βουδαπέστη. Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια παγκόσμια εκστρατεία για τα τουριστικά πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε να είναι μια τηλεοπτική διαφημιστική εκστρατεία σε όλα τα κανάλια που θα παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τουριστικό προορισμό. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Χατζημαρκάκη για να κλείσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους ε, που μου προσέφεραν άλλο ένα κύμα ιδεών. Δεν είχαμε πολύ ε, χώρο για να τα συμπεριλάβω μέχρι τώρα, αλλά θα τα συμπεριλάβω με βάση τις τροπολογίες που έχουν γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία είναι 3 Φεβρουαρίου το μεσημέρι για τις τροπολογίες ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία τώρα ε, παρουσιάσατε να τα δώσετε γραπτό στον κύριο Χατζημαρκάκη για να τα συμπεριλάβει στην έκθεσή του. Και περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του παροπλισμού πυρηνικών σταθμών στα, κράτη, στα νέα κράτη-μέλη. Ο συνάδελφος Μπαλτσίτης είναι ο εισηγητής και του δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πολλοί από τους συναδέλφους μας γνωρίζουν ε, το θέμα αυτό, ο παροπλισμός πυρηνικών σταθμών, πυρηνικών ε, αντιδραστήρων είναι έχει τεράστιες πολιτικ... έχει πολιτικές διαστάσεις και οικονομικές δια... διαστάσεις, ε, κυρίως πολιτικές διαστάσεις. Ε, όπως ξέρετε, οι τρεις κυβερνήσεις ε, από ε, τις διαπραγματεύσεις ε, προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβαν την υποχρέωση να παραπλήσουν τους πυρηνικούς σταθμούς τους. Βεβαίως, ο παραπλησμός κοστίζει και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κονδύλια και στις χώρες αυτές δεν ε, υπήρχαν τα κονδύλια για τον παραπλησμό. Ε, ε, Ελάχιστοι λοιπόν θα πρέπει να ανεβρεθούν από κάπου οι πόροι Γι' αυτό και γι' αυτό νομίζω ότι μέχρι το ότι πρέπει να αναζητηθούν, να, να βοηθήσουμε στην αναζήτηση των πορών αυτών. Μέχρι το 2013 υπάρχουν 2,8 δις. μας κρύψει το 2,8 εκατομμύρια για ε, διαθέσιμα δεν ξέρουμε ε, τι θα γίνει όμως μετά. Το, από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ε, διαπιστώνουμε ότι ε, αρκετά ότι ίσως κάποια κράτη-μέλη δεν χρησιμοποίησαν σωστά τα κονδύλια τα οποία προορίζονταν για τον σκοπό αυτό. Βέβαια θα γίνουν νέες ε, μελέτες και θα υπάρχουν νέα πορίσματα μέχρι το φθινόπωρο του 2011 και πραγματικά περιμένω να δω τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν. Τώρα, από εκεί και πέρα Από εδώ και μπρος βεβαίως προβλέπεται όλοι αυτοί όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί οι οποίοι λειτουργούν να δημιουργούν ένα απόθεμα για τον μελλοντικό του ενδεχομένω παροπλισμό Συγχρόνως θα πρέπει να διατίθενται κονδύλια για την ασφάλεια και δει από εδώ και μπρος αυξημένη ασφάλεια των αντιδραστήρων Πάντως ο παραπλησμός των πυρηνικών σταθμών στις τρεις χώρες ε, αυτές που είναι υποχρεωμένες από το πρωτόκολλο ένταξης να κάνουν κάτι τέτοιο οι τρεις αυτές χώρες θα πρέπει να βοηθηθούν. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος ο κύριος Σουέτσο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική γνωμοδότηση που συνέταξε. Ωστόσο θα είχα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, δεν είναι αλήθεια ότι έγινε πλήρης παροπλισμός των πυρηνικών σταθμών. Ε, για οικονομικό λόγο έλλειψης οικονομικών πόρων δεν, δεν μπόρεσαν να εξυγχρονιστούν οι πυρηνικοί σταθμοί αυτοί. Σε δύο περιπτώσεις, δηλαδή στο Κοσλοντούι υπάρχουν τα προβλήματα αυτά. Οι διεθνείς ε, εμπειρογνώμονες οι οποίοι ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά είπαν ότι θα πρέπει από εκεί και πέρα ό,τι απομείνει να εξυγχρονιστεί αλλά δεν ε, ήταν εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο παντού ε, το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να αναφέρει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά δεύτερη παρατήρηση και οι τρεις χώρες που αναφέρθηκαν ε, σεβάστηκαν τις ανηλυμένες δεσμεύσεις τους χωρίς καμ... να είναι ουσιαστικά προετοιμασμένες ούτε οικονομικά ούτε τεχνικά για να κάνουν κάτι τέτοιο. Και είναι πολύ, ε, είναι νομίζω φυσιολογικό οι χώρες αυτές να ζητούν τη βοήθεια και την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ζητούν να βοηθηθούν στον παροπλισμό των ε, αντιδραστήρων και είναι φυσιολογικό ίσως να γίνουν και κάποια λάθη ή να χρησιμοποιηθούν κάποια ε, κονδύλια όταν πρώτο παρελήφθησαν για μέτρα τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με τον παραπολισμό των πυρηνικών αντιδραστήρων αλλά είναι ενεργειακά μέτρα τα οποία ήταν απαραίτητο να επιβληθούν δεδομένου του παροπλισμού και για να ανταποκριθεί η χώρα στην κατάσταση μετά τον παροπλισμό. Αλλά εγώ νομίζω ότι τα περισσότερα κονδύλια τα κονδύλια στο μεγαλύτερο βαθμό τους χρησιμοποιήθηκαν για τον παραπλησμό των ε, πυρηνικών ενδραστήνων. Και τώρα για την ε, οικονομική βοήθεια που από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η βοήθεια αυτή που δίνεται στις ε, τρεις χώρες ε, δυστυχώς δίνεται κάπως κατακαιρματισμένα. Δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων. Ή υπάρχει έλλειψη συντονισμού για τον οποίο κανείς δεν ενδιαφέρεται. Προβλήματα παραδείγματο χάρη που σχετίζονται με την επεξεργασία ε, ραδιενεργών αποβλήτων η προσέγγι, η, τα προγράμματα αυτά είναι τελείως διαφορετικά στις τρεις χώρες. Αυτό θα μπορούσε να φανταστεί κανείς να γίνεται ε, αν ε, επρόκειται τέλος πάντων πρόκειτο να γίνει μια κάποια σύγκριση μεταξύ αυτών των προγραμμάτων για να επιλεχθούν τελικώς οι βέλτιστες πρακτικές. Ούτε αυτό όμως δεν γίνεται. Λέω λοιπόν ότι η οικονομική βοήθεια που γίνεται στις τρεις χώρες ε, περνάει από το Διεθνές Ταμείο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επενδύσεων. Αλλά οι κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες που απαιτούνται από την τράπεζα δεν είναι οι ίδιοι με τους κανόνες που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο και έτσι δημιουργούνται προβλήματα. Οι διάφορες χώρες αγνοούν τους κανόνες της Τράπεζας Επενδύσεων. η τράπεζα από την άλλη μεριά δεν δέχεται τους εθνικούς κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και στη συνεργασία και στο συντονισμό και στη διαφάνεια κατά τη χρηματοδότηση. Θα κάνω τις σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ ο συνάδελφος Μεσάρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι χώρε αυτέ αναμένουν κάποια χρηματοδότηση ω αντιστάθμιση για τι δαπάνες τι οποίε έχουν καταβάλει οι εργασίες παροπλισμού θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν για να, να υπάρχουν όσο λιγότερες ε, επιπτώσεις είναι δυνατόν. Και θα πρέπει ε, να αναβαθμιστούν εάν ε, είναι δυνατόν οι αντιδρασίες ή να παροπλιστούν εφόσον δεν μπορεί να γίνει αυτό και να, ώστε να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας. Υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις και στο επίπεδο ενεργειακού εφοδιασμού των χωρών αυτών και γι' αυτό θα αναπτυχθούν ε, εναλλακτικοί εναλλακτικές πηγές ε, ενέργειας, πράγμα το οποίο επίσης πρέπει να χρηματοδοτηθεί. και θα παρακολουθούμε τις στρατηγικές που θα εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη αυτά για τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Παράλληλα με τη χρηματοδότηση για τον παροπλισμό των ε, παλαιών πυρηνικών αντιδραστήρων, χρειαζόμαστε και τις δαπάνες για τους νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες, και σε όλες αυτές τις επενδύσεις δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ο στόχος μας είναι η παραγωγή ενέργειας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Yes, uh, thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βαλιάν. Και εγώ χαιρετίζω την έκθεση πρωτοβουλία από την αρμόδια της Επιτροπή. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα ε, σχέδια παροπλισμού, τα οποία διονίζονται και φαίνεται να μην ολοκληρώνονται ε, και να μην υπάρχει κατάλληλος έλεγχος. Παρά το γεγονό ότι γνωρίζω ότι ο παροπλισμό είναι μια αργή ε, διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει και κάποιες δεκαετίες ε, και είναι μια επιχείρηση αυτή καθεαυτή, ε, νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή Ήτρε θα πρέπει να εκφράσουμε και κάποιες ανησυχίες όπως εκφράζει και η Επιτροπή Προϋπολογισμών για να αποστείλουμε ένα στεναρό μήνυμα προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, τα κονδύλια τα οποία διατέθηκαν δεν είχαν ως σκοπό να καλύψουν το πλήρες κόστος του παροπλισμού και να προβλέψουν και όλες τις οικονομικές συνέπειες. Παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι ένα μεγάλο τμήμα αυτών των κονδυλίων πηγαίνουν σε ενεργειακά προγράμματα που θέλουν να αποζημιώσουν για τον παροπλισμό των ε, ε, εγκαταστάσεων αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να επανεξετάσει το ποσοστό των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται για αυτά τα ενεργειακά προγράμματα. Μου φαίνεται κάπως περίεργο το γεγονός ότι τα ενδελεχή προγράμματα παροπλισμού των προγραμμάτων δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και επομένως σε αυτή τη φάση εξακολουθεί να μην υπάρχει ένα ανώτατο όριο ε, ούτε για το κόστος ούτε για τον τρόπο χρηματοδότησης. Επίσης δεν υπάρχει ε, καμία ιδέα για τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες μετά από το 2013 για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να, ε, να λάβουμε ότι ο βασικός στόχος ε, του παραπλησμού των τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι η ασφάλεια. Και ίσως ε, ναι μεν να βιώνουμε χαλεπούς καιρούς αυτή τη στιγμή από οικονομικής πλευράς, αλλά θα πρέπει να επανεστιάσουμε στον πραγματικό στόχο αυτού του παραπλησμού. Ευχαριστώ πολύ. Η απόφαση να διατεθούν κονδύλια για τον παραπλησμό των ε, πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι ορθή. Δυστυχώς, ούτε όταν λήφθη απόφαση, ούτε όταν ε, ε, ξεκίνησε η διαδικασία για, για το πρώτο εργοστάσιο δεν υπήρχε κάποια προθεσμία και κάποιο ανώτατο όριο προς το κόστος και τη λήξη του. Δεν ξέρει λοιπόν κανείς πότε θα περατωθεί η διαδικασία ούτε ποιο θα είναι το συνολικό κόστος. Όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως έχουν δαπανεθεί πάρα πολλά χρήματα σε ε, ενεργειακά προγράμματα τα οποία περιλαμβάνονται σε επιλέξιμες δαπάνες. Από πλευρά Επιτροπής μας θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον τα όσα, έχουν γίνει για τα ενεργειακά αυτά προγράμματα μέχρι τούδε έχουν καλύψει τις απώλειες οι οποίες έχουν προκύψει από τον παροπλισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Εάν θεωρούμε ότι χρειάζονται περαιτέρω επενδύσει σε ενεργειακά προγράμματα, τότε θα πρέπει να υπάρξει μια ομάδα συντονισμού, μια ομάδα καθοδήγησης, προκειμένου να καθοριστεί το κόστος. Και επίσης χρειάζεται ένα διεξοδικό σχέδιο για να γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, ποιο είναι το συνολικό κόστος και ποια είναι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το κόστος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Οντή. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα έργα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ νομίζω ότι ανέφερε ο συνάδελφος και σε μια προηγούμενη έκθεση για τον πυρηνικό σταθμό του Κόσλοντούι το είχαμε αναφέρει, να μπει μια ρήτρα κοινοτική προτίμηση. γιατί υπάρχει τεχνογνωσία στην Ευρώπη για τέτοιες εργασίε παροπλισμού πυρηνικών σταθμών. Από τις, ε, τα δημόσια αυτά κονδύλια δεν μπορούμε να έχουμε δημόσιες συμβάσεις που θα δίνουν τα έργα αυτά σε εταιρείε τρίτων χωρών χωρίς να προσφέρουν την ευκαιρία και στις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Να βάλουμε λοιπόν μια ρήτρα κοινοτικής προτίμησης σε, αυτέ τι αυτές τις συμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους και για την ανταλλαγή απόψεων. Όταν μίλησα για το θέμα αυτό και μάλιστα αν είχα περισσότερο χρόνο για να πω περισσότερα, θα μπορούσα να σας πω πολλά και πάλι δεν θα ήταν αρκετά για μια καλή γνωμοδότηση, θα, είχα, θα έπρεπε να μακρηγορήσω. Θα μπορούσα να μιλήσω και για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και αυτό που είπε ο κύριος Σοντή είναι χρήσιμη παρατήρηση. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση και για τις ιδέες ε, που συνεισφέρατε. Ο παροπλισμός των πυρηνικών αντιδραστήρων πρέπει να ολοκληρωθεί και πρέπει να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια. Και το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του θα δείξει αν απαιτείται κάποια ομάδα μελέτης επί, του, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πόσο κοστίζει η νέα κατασκευή ενός νέου πυρηνικού αντιδραστήρα και να συνυπολογίσουμε τον παροπλισμό καθώς και το κόστος διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων γιατί μπορεί να καταλήξουμε τελικά σε εντελώς διαφορετικά ποσά και να δούμε ε, το αν η πυρηνική ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας που δεν είναι τόσο δαπανηρή όσο πολλοί ισχυρίζονται. Νομίζω ότι με αυτή την έκθεση θα προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα που θα μας απασχολήσουν για μελλοντικέ περιπτώσεις παροπλήσμου πυρονικών αντιδραστήρων. Αν δεν υπάρχει ε, άλλο σχόλιο, ε, θα ήθελα να σας πω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι το μεσημέρι στις 3 Φεβρουαρίου. Και περνάμε στο σημείο 8 μέθοδη πρόσβαση στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Ραδιοπλοήγηση που προέκυψε από το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεση και δίνω το λόγο στον συνάδελφο Γκλάντε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω ότι όλο και λιγότεροι γινόμαστε. Δεν ενδιαφέρονται και πολύ για το θέμα αυτό, γιατί θα, γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομος. Το Γαλιλαίο τελικά και το σχετικό πρόγραμμα προσφέρει πέντε υπηρεσίες. Ε, ανιστιχτή υπηρεσία, εμπορική υπηρεσία, ασφαλή υπηρεσία, υπηρεσία αναζήτηση και διάθεση και την κυβερνητική υπηρεσία PRS για την οποία θα μιλήσω εγώ τώρα. Ε, πρόκειται για μια υπηρεσία την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, και οι εθνικές κυβερνήσεις για την πυροσβεστική, για την αστυνομία και τα λοιπά, αλλά και ε, άλλες και το Συμβούλιο και η Επιτροπή και τα λοιπά αυτά προβλέπονται στο πλαίσιο που της πρότασης στο πλαίσιο που προτείνεται προτείνονται Προτείνονται επίσης ε, μέθοδοι εποπτείας και προτείνονται και ε, διαδικασίες αδειοδότησης των χρηστών. Εδώ γιατί τα αντικείμενα που πραγματεύεται τελικά αυτό το, αυτή η υπηρεσία, με την οποία ασχολείται αυτή η υπηρεσία είναι αρκετά ευαίσθητα. Ε, ε, ε, χρειάζεται λοιπόν, χρειάζεται μεγάλη εποπτεία και έλεγχος λοιπόν. Τώρα τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί μπορούν να, να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή αν και εφόσον υπογράψουν κάποιο συμφωνητικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρόταση λέγεται παρακάτω, λέγεται επιπλέον ότι Ε, θα πρέπει να καθοριστούν ε, οι προϋποθέσεις που τις οποίες χρησιμοποιείται η υπηρεσία αυτή, να καθοριστούν αυστηροί κανόνες ε, και εγώ θα ήθελα να πω ότι θεωρώ την πρόταση αυτή αρκετά ικανοποιητική. Το υπηρεσία αυτή είναι μια από τις βασικές υπηρεσίες προσφέρεται από τον Καλλιλέο. Ε, Υπάρχει βεβαίως ο κανονισμός Γαλιλαίο με τους ε, συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες ε, και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτές τις διαδικασίες για να πάμε παραπέρα. Για την ασφάλεια τώρα του, του, του συστήματος θα πρέπει να οριστούν κάποιες εθνικές αρμόδιες αρχές. Εάν οι αρχές αυτές δεν ε, μπορούν να ανταποκριθούν, τότε παρεμβαίνει η Ένωση και ε, αναλαμβάνει και ε, βοηθάει κατά κάποιο τρόπο ή αναλαμβάνει, βοηθάει στην αναλαμβάνει την εποπτεία, βοηθάει στον έλεγχο. Ε, από εκεί και πέρα βεβαίως, ιδιαίτερα με τις τρίτες χώρες, τα προβλήματα είναι ε, αρκετά σημαντικά. Όλοι ξέρουμε τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τον Γαλιλαίο. Ξέρουμε τις δυσκολίες λοιπόν που αντιμετωπίσαμε και δεν θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε αντίστοιχε ε, δυσκολίες στο μέλλον. Δεν ξέρουμε επίσης τι θα γίνει με τους Κινέζους. Αυτά εντός παρενθέσεως. Ε, πάντως ε, θα υπάρχουν κανόνες, πρέπει να υπάρχουν κανόνες, πρέπει να εποπτεύεται η συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανόνες ασφαλείας προ, προφανώς. Τώρα για τη, χρηματοδότηση ή το κόστος του, της υπηρεσίας αυτής, το δεν θα καταβάλλεται από τους χρήστες αλλά από τους συμμετέχοντες και φανταζόμαστε εδώ ο, εταιρικές σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ε, ε από εκεί και πέρα περιμένω τις ιδέες σας μέχρι τις 2-3 ε, Φεβρουαρίου. Ξέρω ότι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έγινε μια αρκετά έντονη, ζωντανή συζήτηση για το θέμα αυτό. Ε, ευχαριστώ για την υπομονή Ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι η εκθέση του κύριου Γκλάντε είναι πολύ τεχνική και γνωρίζω ότι μπορούμε ακόμα να κάνουμε κάποιες μικρές αλλαγές. Ιδίως όταν μιλάμε για χρηματοδότηση θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία από πλευράς μας ότι τόσο από πλευράς λειτουργικότητας, ιδίω για το σύστημα PRS, θα πρέπει να συνεχίσει όλη η διαδικασία, διότι ε, μας δίνει πολύ περισσότερα από το σύστημα GPS και επίσης ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, θα πρέπει ε, να ξεχάσουμε τις παραδοσιακές μεθόδους χρηματοδότησης. Διότι θα έχουμε καλά ωφέλη, ιδίω για χώρες οι οποίες θα λάβουν το βάρος ε, του προγράμματος αυτού. Από τις τροπολογίες διαπιστώνω ότι κάνετε μία απόπειρα να βρείτε την κατάλληλη ισορροπία Απ' τη μια υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά από την άλλη υπάρχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίε οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε δύσκολη ε, κατάσταση και μπορεί να μην θέλουν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση. Αυτό αντικατοπτρίζεται σαφώς στις τροπολογίες. Όπως είπατε κι εσείς, ε, μπορώ να ακολουθήσω τις ε, τροπολογίες σας. πρέπει να υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης. σαφώς είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο πιο επισταμμένα. Δεν έχω καμία αμφιβολία από αυτού. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερο τεχνικό, αλλά αν δεν μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά μακροπρόθεσμα και αν το κερασάκι στην τούρτα δεν το χρησιμοποιήσουμε εμείς, δεν το βάλουμε εμείς, μάλλον θα μας εξαφανίσει το πεντάγωνο, θα μας υποχρεώσει να χαθούμε από το προσκήνιο. Καλό λοιπόν θα ήταν να έχουμε τέτοιες τροπολογίες. Να πω όμως ότι υποστηρίζω πλήρως αυτά τα οποία ε, ε προσπαθείτε να εξισορροπήσετε. Ευχαριστώ η κυρία Χολ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τα όσα κάνατε και να ρωτήσω κάποια διευκρινιστικά στοιχεία για να είμαι βέβαιη ότι κατάλαβα καλά. Μας λέτε ότι όσον αφορά το κόστος, τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν θα πρέπει να είναι αυτά τα οποία πληρώνουν και από εκεί και πέρα τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν πώς θα ανακτήσουν αυτό το κόστος από τους χρήστες. Ορθώς κατάλαβα. Ωραία, ευχαριστώ. Συνάδελφος ε, Ρέμεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο εισηγητής ε, και εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο που έχει κάνει. Είναι άλλο ένα σωστό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι πρέπει να το δούμε. Δεν έχω πρόβλημα με τα περισσότερα θέματα που υπάρχουν μέσα στο κείμενο αυτό. Θα τα υποστηρίξω. Είναι ένα πολύ τεχνικό θέμα. Αλλά δεν είναι και 100% τεχνικό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει ο εισηγητής στο τέλος. Ότι θα πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε. Είναι ένας νέος τομέας στον οποίο δεν έχουμε πείρα και θα πρέπει να διαμορφώσουμε τους κανόνες. Εδώ μιλάμε για συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Και νομίζω ότι η παρούσα ευκαιρία είναι πολύ καλή γιατί είναι μια απόφαση που προήλθε από την ε, συνεδρίαση του αρμόδιου οργανισμού και νομίζω ότι προχωράμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με αυτούς που ε, συνεχάρισαν και θεώρησαν θετική τη δουλειά που έκανε ο κύριος Γκλάντε. προώθησε όλη αυτή την υπόθεση ένα βήμα ακόμη ο κύριος Γκλάντε και εδώ θα πρέπει να είμαστε όλοι ανοιχτοί. Θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι διότι η τεχνολογία είναι ρευστή και αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά σε μερικά χρόνια μπορεί αυτά τα οποία συζητάμε εδώ είναι ήδη πεπαλαιωμένα, είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, αυτά που λέει ο κύριος Γκλάντε και ειδικά για την κυβερνητική υπηρεσία, PRS. Ε, τα πράγματα είναι πολύπλοκα, υπάρχουν οικονομικά ε, έντονες οικονομικές διαστάσεις εδώ και βεβαίως ε, όλα αυτά σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του Γαλιλαίου, αλλά ευτυχώ βρισκόμαστε στον πολιτικό τομέα εμεί. Δεν είμαστε στα, στο GPS όπως οι Αμερικάνοι, οι οποίοι στηρίζονται στρατιωτικό τομέα για το χρηματοδότηση του GPS. Εν πάση περιπτώσει χαίρομαι ιδιαίτερα που α, έκανε τη γνωμοδότηση αυτή ο κύριος Γκλάντε και ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ε, όχι μόνο για τη χρηματοδότηση του PRS αλλά και για την ε, παροχή κονδυλίων για την εγγύηση της ασφάλειας στο σύστημα ε, στην υπηρεσία αυτή. Υποστηρίζω λοιπόν τη γνωμοδότηση αυτή γιατί πιστεύω πως πρόκειται για ένα σοβαρότατο ζήτημα που περιλαμβάνει οικονομικές, ε, πολιτικές, νομικές πτυχές. Ευχαριστώ τον κύριο Κλάντε για τη δουλειά που έκανε και προσβλέπω στις μελλοντικές συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ, ο πρόεδρος, ο κύριος Μπόσκος, ζήτησε το λόγο. Θέλετε το λόγο ή... Παρακαλώ. Euh. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε συγητά, κυρίες και κύριοι. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη θετική αντιμετώπιση της πρότασης ε, της ε, Επιτροπής. Και ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατόν η συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα κείμενο που θα εγκριθεί τον Ιούνιο. Θέλησα να λάβω το λόγο για να προλάβω μελλοντικέ συζητήσεις όταν θα συζητηθούν οι τροπολογίες και θα είμαι σύντομος. Στις ε, τροπολογίες ε, σημείωσα κάποια θέματα που αναφέρονται που έχουν σχέση με τη σαφήνεια των ορισμών Υπάρχει η έννοια του χρήστη και του ε, αδειοδοτημένου χρήστη. Participants και users στα αγγλικά. Θα χρειαστεί κάποιο κείμενο ορισμών. Θα συντάξουμε λοιπόν τους ορισμούς για να μην υπάρχει αμφισημία στο κείμενο για τους όρους που χρησιμοποιούνται. Το θέμα της ανάληψης του λειτουργικού κόστους επίσης ε, είναι σημαντικό για τη χρήση της κυβερνητικής υπηρεσίας. Όπως λέει και η έκθεση, έτσι και η Επιτροπή πιστεύει ότι τα κράτη-μέλη και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί που συμμετέχουν θα πρέπει να είναι αυτοί που φέρουν το λειτουργικό κόστος. Παρ' όλα αυτά, ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να επιλέξουν ε, τη μετακύληση του κόστους ή τμήματος του κόστους στους τελικούς χρήστες. Μιλάμε για ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως. Μιλάμε για 100.000 ευρώ περίπου. Ε, δεν θα έλεγα ότι είναι δυσβάστακτο το κόστος αυτό για το κράτος μέλος και για τους τελικούς χρήστες. Και στην έκθεση αλλά και στις παρεμβάσεις ε, των μελών της Επιτροπής σημείωσα ότι προέκυψε το ερώτημα του ρόλου των τρίτων χωρών στη χρήση της κυβερνητικής υπηρεσίας ή στην κατασκευή των δεκτών PRS. Όσοι έχει τώρα το κείμενο, ως λύση αναφέρεται μια ενδεχόμενη διεθνής συμφωνία και κάτι τέτοιο θα δώσει την απαραίτητη ευελιξία ώστε κατά περίπτωση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των τρίτων χωρών. και θα είμαστε ανοιχτοί για να υποβάλουμε τις κατάλληλες προτάσεις κειμένου για να διευκρινίσουμε τις συγκεκριμένες παραγράφους της αιτιολογικής έκθεσης. Μια τελευταία παρατήρηση. για την πρόταση της διαδικασίας που υπάρχει λεπτομερώς μάλιστα για τα στάδια της διαδικασίας που θα εφαρμοστούν αν δεν τηρηθούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που θα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων στην κυβερνητική υπηρεσία. Προτείνονται κάποιες λεπτομέρειες που τις βρίσκουμε ιδιαίτερα σωστές και νομίζω ότι θα είναι σκόπιμο να ενταχθούν στο κείμενο. και θα αποτελέσουν το βασικό άξονα αυτών τα οποία στη συνέχεια θα εγκριθούν. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σημειώνω ότι πολλοί βουλευτές μίλησαν υπέρ μιας συμπληρωματικής χρηματοδότησης. Κάτι με το οποίο συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Κύριε και πάλι για τη χρηματοδότηση Κοιτάξτε να δείτε, η χρηματοδότηση πάει στα, ε, την αναλαμβάνει από εκεί και πέρα ε, το, την επιστροφή αν θέλετε της χρηματοδότησης την κανονίζουν τα κράτη-μέλη θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα για την πυροσβεστική όπως σας είπα για την αστυνομία κτλ οπότε θα δουν εκείνοι από εκεί και πέρα τι θα γίνει και από εκεί και πέρα βεβαίως ε, δεν είμαι σίγουρος ότι θα, η χρηματοδότηση έτσι όπως τη φαντάζομαι θα λειτουργήσει θα περιμένουμε να δούμε, θα δούμε και τις τροπολογίες ναι λέει ο πρόεδρος δεύτερη 2 Φεβρουαρίου 12 η ώρα το μεσημέρι η ημερομηνία για την κατάθεση των τροπολογιών και τώρα πάμε στο επόμενο θέμα τη σημερινή διάρκεια, το παλιό 6 Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ευρυζωνικότητας επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη. Η συγγήτρια είναι η κυρία Τζαβέλα, στην οποία και δίνω αμέσω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας έχω ήδη διανύμει ένα τυπο έγγραφο εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει κάποιες από τις προτάσεις μας για ε, τα ευρωπαϊκά ευρυζωνικά δίκτυα. Καταρχάς να σας πω ότι το κόστος της μη ψηφιακής Ευρώπης είναι πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κερδίσει ένα 4% του ΑΕΠ εάν ε, δώσει την αίθουσα για την πρώτη ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς μέχρι το 2020. Αυτό αντιστοιχεί σε κέρδος περίπου 500 δις ευρώ. Ω προ την έκθεση τώρα, κατά την άποψή μου, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το 2020 καθαρίζονται κατά τρόπον ώστε τα ωφέλη αλλά και τα μειονεκτήματα θα αρχίσουν να φαίνονται μακροπρόθεσμα. Είναι πολύ καλή η στόχη, τους ε, ε, χαιρετίζω και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τις προτάσεις της. Σε αυτή την έκθεση θεωρώ ότι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούμε είναι το βασικό, ο βασικός στόχος ευρυζωνικού δικτύου για το 2013 που είναι να έχουμε 100% κάλυψη ευρυζωνικού δικτύου στους πολίτες των 27 κρατών μελών. Εξού και στο σημείο 5 του εγγράφου εργασίας αναφέρω ότι ο στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι να έχουμε ε, παγκοσμίω τον ηγετικό ρόλο σε υποδομές πληροφορικής και επικοινωνίας μέχρι το 2013, ε, παραδίδοντας ε, περίπου 100% κάλυψη σε ευρυζωνικό δίκτυο, δίνοντας ε, τουλάχιστον 2 Mbps ε, σε κάθε χρήστη. Θεωρώ ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός και για τα 27 κράτη-μέλη και πρόκειται για ένα στόχο ο οποίος μπορεί να επιτευθεί στο εγγύς μέλλον. κατά αυτόν τον τρόπο εστιάζουμε σε βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους. Επιπλέον, είναι υψής της σημασίας να σημειώσουμε ότι η πρόσβαση 100% σε ευρωζωνικό δίκτυο και το να υπάρχει δυνατότητα για 100% ευρωζωνικό δίκτυο θα είναι ε, χαμένος σκόπος εάν δεν συμπεριλάβουμε μία στεναρή στρατηγική για να διασφαλίσουμε ασφάλεια του κυβερνοχώρου και ε, διαδικτυακή ασφάλεια. Ένα ακόμα θέμα που μας απασχολεί στην έκθεση αυτή και σαφώς θα πρέπει να το αναφέρουμε έχει να κάνει με την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές ε, και νήσους. Θα πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα ώστε οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στους τομείς αυτούς και θα πρέπει να επισημάνουμε την ανάγκη να ε, χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις συμπληρωματικές τεχνολογίες προκειμένου να έχουμε ευρυζωνική κάλυψη σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές χωρίς να υπάρχει ε, επιπλέον άχθος για τις επιχειρήσεις και τους ε, καταναλωτές. Κατά αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι οι οπτικές ίνες θα πρέπει να είναι η βασική πλατφόρμα για να παρέχουμε τα 100 MB και πρέπει να σκεφτούμε και τη χρήση και την πρακτική εφαρμογή και άλλων, και άλλων μορφών πλατφόρμας όπως για παράδειγμα ε, των δορυφορικών. Πρόκειται για πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν και να μπορέσουμε να παρέχουμε ευρυζωνικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες ε, και ε, περιοχές και περιοχές της υπαίθρου. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε πόσο σημαντική είναι να υπάρχει κατάλληλη κατανομή του φάσματος για ε, ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της χρηματοδίτησης. Οι πρόσφατες στατιστικές μελέτες μας δείχνουν ότι οι στόχοι για το 2010 ήταν τετραπλάσιοι από το 2009 και είχαμε 1,8 δις από δημόσιους πόρους, ε, ποσό ρεκόρ. Θεωρώ λοιπόν ότι η στοχευμένη χρήση κοινοτικών πόρων και η συγκεκριμένη κρατική επιδότηση για την ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι η βασική πηγή για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την ευρυζωνική διάθεση. Επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ε, δίκτυο και να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι και η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών αλλά και της κεντρικής κυβέρνησης για τους στόχους επενδύσεων για τις τηλεπικοινωνίες. Πριν ολοκληρώσω θα ήθελα επίσης να ζητήσω και να εκφράσω την υποστήριξή μου για τη δημιουργία μιας ομάδας ειδικών καθητών υψηλού επίπεδου για να μπορέσουμε να έχουμε μελλοντικές ε, ε, στρατηγικές για υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών. Η πληροφορική και επικοινωνίες είναι ένας τομέας ο οποίος κινείται ταχύτατα και επομένως θα πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να εξεύρουμε κοινέ λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται ε, με προεξάρχοντα ρόλο στα θέματα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Η ανάπτυξη αυτή θα μας δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τον κύριο κινητήριο μοχλό μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής ατζέντα και της μετατροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ψηφιακή οικονομία. Προσβλέπω στη συνεργασία με τους συναδέλφους από όλες τις ομάδες εργασί... Ε, πολιτικές ομάδες συγγνώμη, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα μας οδηγήσει στη νέα εποχή εποχή, την ψηφιακή εποχή και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνδρομή της και την υποστήριξή της για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mr. Um Chairman. I, I will do as well in English. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα τα πω αγγλικά για να μην καθυστερούμε και να ξεκουρασώ λίγο και τους διερμηνείς, λέει ο, ο μιλητής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, διότι μας έδωσε μια καλή βάση για συζήτηση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Αφενός, όπως και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, έτσι και το σχέδιο κειμένου σας, είναι ισορροπημένο και καλύπτει όλα τα βασικά στοιχεία. Κατά κάποιον τρόπο όλα είναι σαφή. Δεν βρίσκουμε κάποιο πτέσμα. υπάρχουν όλα τα στοιχεία που αφορούν την ψηφιακή ατζέντα και ούτε καθεξής. Από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες στις οποίες θα πρέπει να σταθούμε και τις οποίες θα πρέπει να επισημάνουμε. Είμαι υπέρ του γεγονότος ε, ότι θα πρέπει να έχουμε αυτούς τους στόχους, τους βραχυπρόθεσμους για το 2013 για 100% κάλυψη και τουλάχιστον 2 Mbps. Αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα έπρεπε ίσως να τονίσουμε στην έκθεσή σας. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε δύο τομείς. Ε, to come back to your previous να σας παραπέμψω στο προηγούμενο εγγραφό σας, στο οποίο αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στις πρωτοβουλίες. Ίσως θα έπρεπε να επανέλθετε στο σκήμενο αυτό και να το επεκτείνετε λίγο, διότι η ηλεκτρονική υγεία, για παράδειγμα, και άλλοι τομείς, οι οποίοι χρειάζονται ε, κατάλληλη διαχείριση αλλά και ε, προσέγγιση από πλευράς αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων θα μπορέσουν ίσως να μας δώσουν νέους τομείς για ιδιωτικές δραστηριότητες και επενδύσεις. Μια δεύτερη παρατήρηση για το σλόγγαν που χρησιμοποιείτε, το Broadband for All. για να έχουν ευρυζωνικέ υπηρεσίε όλοι, χρειαζόμαστε κατάλληλε υποδομέ, χρειαζόμαστε τι επενδύσει και την οικονομική προσέγγιση, αλλά κάποια αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν και τα έχω από τη χώρα μου τη Λιθουανία. Δεν θα αρχίσω τώρα να σας απαριθμώ τα στοιχεία, αλλά όπως αποδεικνύεται και από τα δικά σα τα στοιχεία, στη Λιθουανία η κάλυψη του ADSL είναι ήδη στο 80% και κατά πάσα πιθανότητα θα καταφέρουμε να τηρήσουμε το στόχο. Από την άλλη, το ίντερνετ εξαρτάται πάρα πολύ από το εισοδήματο και έχουμε στοιχεία για τα νοικοκυριά. Αν δούμε δηλαδή τα πλουσιότερα νοικοκυριά, εκεί έχουμε κάλυψη κατά 95% και αυτοί που λαμβάνουν το 1 τρίτο των άλλων νοικοκυριών έχουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό χρήση. Είναι και κοινωνικό λοιπόν το φαινόμενο, υπάρχει κοινωνική πτυχή και νομίζω ότι θα πρέπει να τη σκεφτούμε για το μέλλον. Ίσως θα μπορούσαμε να ε, έχουμε και αντίστοιχα παραδείγματα από άλλες χώρες. Αυτά ως πρώτη εντύπωση. Να συγχαρώ για άλλη μια φορά την εισηγήτρια και Επειδή είμαι σκιώδης εισηγητής ε, για το ΕΛΚ, ε, θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση και περιμένω να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Η κυρία Βάλεα, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι έχουμε μια ισορροπημένη πρόταση. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί για τους ε, στόχους που θέτουμε για την ψηφιακή ατζέντα θα πρέπει να έχουμε και τα μέσα για να τους επιτύχουμε και από ό,τι φαίνεται από αυτή την ανακοίνωση έχουμε ένα πρώτο θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους φιλόδοξους στόχους για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και να έχουμε περαιτέρω υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικό ε, διαδίκτυο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τις άλλες οικονομίες. Το διαδίκτυο είναι στον πυρήνα της κοινωνίας μας ε, σε πολλούς τομείς, ε, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στην άμενα, στην καθημερινή μας ζωή και η ανάπτυξη γρήγορων ευρυζωνικών δικτύων είναι απαραίτητα και για τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις για να υποφεληθούν της ψηφιακής οικονομίας και να ανταποκριθούν στις ε, ε, ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες για βελτιωμένες υπηρεσίες. Να σας πω ποιες θεωρώ εγώ προτεραιότητες. Καταρχάς, θεωρώ ότι ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον και τα καλύτερα κίνητρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις στις υποδομές ευρυζωνικών δικτύων και γι' αυτό το σκοπό θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ανταγωνιστικές ευρυζωνικές αγορές. Επειδή οι επιλογές των καταναλωτών είναι ίσως ο πιο βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη υψηλή ταχύτητας ευρυζωνικού δικτύου στην Ευρώπη, ε, θα πρέπει οι εθνικοί ρυθμιστές να να εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όταν αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός ε, και της παροχής υπηρεσιών και των υποδομών και ε, να μην υπάρχει διάκριση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Και εδώ δεν αναφέρομαι μόνο στον ανταγωνισμό των υπηρεσιών και στην ε, δίκαιη πρόσβαση, αλλά και στον ανταγωνισμό μεταξύ των υποδομών ως σημαντική πτυχή για τις επενδύσεις. Οι οπτικές ίνες και το κινητό ευρυζωνικό δίκτυο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν. Δεύτερον, σε τομεί στου οποίους δεν είναι οικονομικά βιώσιμες οι ιδιωτικέ επενδύσεις, θα πρέπει να γίνουν δημόσιες επενδύσει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει, τίθεται πλέον το ερώτημα. Θα πρέπει να υπάρχουν δημόσιες διαπάνες ε, όπου οι ιδιωτικέ επενδύσεις δεν επαρκούν. Ενώ η έκθεση αυτή ε, μιλά για περισσότερε ιδιωτικέ επενδύσει για μείωση του κόστου και ε, την αύξηση τη νομική σαφήνεια η σωστή χρήση και ο συντονισμός των ε, διαρθρωτικών ε, ταμείων και του Ταμείου Ανάπτυξης της Υπέρθης, ε, Υπέθρου θα δημιουργήσουν συνέργειες για τα προγράμματα υποδομών. Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στις ε, τρέχουσες τάσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα αυτών των τάσεων. Θα πρέπει να έχουμε σαφείς μετρήσιμους στόχους μέσω κατάλληλων δικτών και ε, θα πρέπει τα κονδύλια να δαπανούνται καταλήλως να υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο εποπτείας και κατάλληλος έλεγχος από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προγράμματα που εφαρμόζουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Χαιρετίζω επίσης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να συμμετέχει πιο ενεργά στη χρηματοδότηση του ευρυζωνικού δικτύου για να συνάδει και με τους στόχους της Ευρώπης του 2020 που θεωρώ ότι θα έχει πολύ καλή επίδραση και σε άλλες τράπεζες. Θα έχουμε και άλλα κονδύλια για το ευρωζωνικό δίκτυο. Επίσης είμαι υπέρ της δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών μέσων, όχι απαραίτητο νέων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ή να επαναχρησιμοποιήσουμε χρηματοδοτικό μέσο για να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα ευρυζωνικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα εγγύησης δανείων, και θεωρώ ότι αυτά είναι βασικά βήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και προσβλέπω στην μελλοντική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας πω για άλλη μια φορά ότι όλοι οι δημόσιες επενδύσεις και τα προτιμησιακά δάνεια θα πρέπει να δίνονται για ε, υποδομές οι οποίες θα υποστηρίξουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των υπηρεσιών και τη δυνατότητα να επιλέξουν καταναλωτές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεάντζελης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ταχεία και ταχύτατη πρόσβαση του διαδικτύου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, όπως έγινε τον καιρό του και με τις μεταφορές και την ηλεκτρική ενέργεια. Αφετέρου, η ανάπτυξη του ευρυζωνικού δικτύου είναι από τους βασικούς πυλώνες της ε, ψηφιακής ατζέντα και αποτελεί πρωτοβουλία φάρο για την Ευρώπη του 2020 για μια ευφυή, βιώσιμη, ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει τους πάντες. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, πολύ καλή δουλειά της, η οποία ήταν και διδακτικής φύσεως, ιδίως όσον αφορά κάποιες ε, θετικές πτυχές. Αναφερθήκατε στην ανάπτυξη των νέων δικτύων. Θεωρώ ότι οι ίσες συνθήκες πρόσβασης στην αγορά των τηλεπικοινωνιών είναι μία αρχή την οποία θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε παντού και πάντοτε. Γι' αυτό ακριβώς και κάνω μία έκκληση ώστε αυτό το σχέδιο έκθεσης να περιλαμβάνει και κάποια επιπλέον στοιχεία για την ανάγκη να καθορίσουμε ισότιμες συνθήκες για την πρόσβαση στα δίκτυα. Μας ενδιαφέρει επίσης να ενισχύσουμε τις υποχρεώσεις ε, κοινών υποδομών προκειμένου να ε, αναπτυχθούν οι επενδύσεις ένα τελευταίο σημείο. Επειδή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η Ευρώπη αποφασίζει να επενδύσει ενεργά σε κάθε σπίτι, σε κάθε επιχείρηση, σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, που σημαίνει ότι θα έχουμε ανάπτυξη και καινοτομία, θεωρώ λοιπόν ότι η σταδιακή αύξηση των μηνιαίων ε, τιμών που θα οφείλονται σε συντήρηση των ε, ε, δικτύων που προηγουμένω ήταν μονοπόλιο θα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικό. Σας το λέω αυτό διότι αν η Ευρώπη πραγματικά θέλει μέχρι το 2020 να έχει ταχύτητες σύνδεσης που θα είναι άνω των 30 MB ανά δευτερόλεπτο και θα είναι διαθέσιμες για όλους τους Ευρωπαίους πελίτες το κατεπηγόντος στην Ευρώπη να υπερισχύσουν τα επιχειρήματα επιχειρήματα των καταναλωτών και να έχουμε μια αγορά η οποία θα είναι ανοιχτή προς όλους και ε, ανταγωνιστική. Η κυρία Δελκαστήγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια, την ε, κυρία Τζαβέλα, για αυτή την ε, ε, παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέσουμε το πλαίσιο αυτού του εγγράφου για την ανάπτυξη του ευρυζωνικού δικτύου στο πακέτο για το ευρυζωνικό δίκτυο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουσιαστικά έχουμε τρεις πρωτοβουλίες. Η μία πρωτοβουλία έχει να κάνει με το φάσμα, η δεύτερη έχει να κάνει με τη σύσταση που έγινε για την πρόσφαση σε δίκτυα νέας γενναίας και η τρίτη είναι αυτή που αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στο ευρυζωνικό δίκτυο θεωρώ ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε εκ παραλίλου με το φάσμα και την πρόταση για το φάσμα που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα το συζητήσουμε άλλωστε. Υπάρχει το έγγραφο εργασίας για το θέμα αυτό του συναδέλφου Χόπμαν και θεωρώ ότι πολύ ορθώς έπραξε η εισηγήτρια επισημένοντας τη σημασία που έχει το φάσμα βάσει και των όσων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι θα πρέπει να καλύψουμε όλες τις πτυχές και όλες τις απαιτήσεις για την απελευθέρωση ε, των 800 MHz και φυσικά και άλλες ε, προτάσεις που θα μας κάνει ο εισηγητής του φάσματος και που έχουμε συζητήσει σε διάφορες περιπτώσεις. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται κατά την έποψή μου και δεν θα πρέπει να λησμονούμε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ψηφιακή ατζέντα να έχουμε ως στόχο όλα οι κατοικίε να έχουν για το 2020 μια ευρυζωνική σύνδεση με πρόσβαση 30 MB και το 50% των κατοικιών για το 2050 να έχουν πρόσβαση με ταχύτητα 100 MB. Μπορεί να φαίνεται σε κάποιους ότι κάνουμε μια πρόταση χωρίς νόημα επενδύσεις αυτή τη στιγμή και πολύ φιλόδοξους στόχους για αυτά τα οποία απαιτούνται. Είναι αλήθεια ότι σήμερα ακόμα και αυτοί που κάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή κατανάλωση στο διαδίκτυο δεν χρειάζονται ταχύτητα που να επιτρέπει 100 ε, MB. Αλλά τα πάντα προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα. Και όταν θα εφαρμόσουμε όλες αυτές ε, τις ε, τεχνολογίες και τα μέτρα που συζητάμε, η στόχη αυτή θα είναι πραγματικότητα και θα βρισκόμαστε πολύ πιο κοντά σε μια ανάπτυξη του διαδικτύου, η οποία θα αφορά πολύ περισσότερες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Ε, είναι αυτό που αποκαλούμε το διαδίκτυο των πραγμάτων. Για όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα χρειαζόμαστε ταχύτητες ε, αυτής της μορφής και επειδή θα πρέπει να υπάρχει μία μακροπρόθεσμη προοπτική που στην πραγματικότητα είναι πολύ βραχυπρόθεσμη θα πρέπει να υπάρχει φιλοδοξία όπως φαίνεται και στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να περιλαμβάνεται δηλαδή εδώ και η ανάγκη να φτάσουμε στο μέλλον σε αυτές τις ταχύτητες. Ευχαριστώ. Να προσέξουμε να μην αργήσουμε. Ο κύριος Κάλφιν ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όπως έκανε και η συνάδελφή μου την κυρία Τζαβάρα για το έγγραφό της είναι μια πολύ καλή βάση για συζήτηση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η πολιτική μας ομάδα των σοσιαλιστών θα υποστηρίξει οτιδήποτε που θα μας οδηγήσει σε γρήγορη ανάπτυξη της ψηφιακής ατζέντα και των νέων τεχνολογιών. Θα θέλαμε, μια και έγινε, και έγινε και λόγος για τις υποδομές και τη χρήση του ίντερνετ, θα θέλαμε να αναφέρουμε κάποια θέματα ε, να αναφέρουμε και ορισμένα σημεία τα οποία εμεί απασχολούν ε, πολύ εδώ στο Κοινοβούλιο. Παραδείγματο χάρη την καθολική κάλυψη uh, και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει πρόσβαση όλος ο κόσμος. Βεβαίως οι υποδομές είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το αναφέρει και η κυρία Τζεβέλα. Το θέμα είναι να δούμε, είναι αλήθεια αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε και όλες ποιες είναι οι υπηρεσίες που θα προκύπτουν από αυτή την υποδομή. Υποστηρίζω τις προτάσεις που κάνει η, η συγγήτρια uh, like... για την ασφάλεια στην κυβερνο, στον κυβερνοχώρο είναι ένα σοβαρότερο θέμα που πρέπει βεβαίως να το λάβουμε υπόψη μας και δεν πρέπει να μελήσουμε την πτυχή αυτή κατά την προσπάθεια μας να διευρύνουμε τις ευρυζωνικές συνδέσεις. Τώρα, έγινε μια κάνατε μια πρόταση να δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα εργασίας, μια task force για να ασχοληθεί με τα συναφή θέματα. Ναι, δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά ε, ε, εκείνο που είναι σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να συνειδητοποιήσουν, να ξέρουν ακριβώς ε, περί τίνος πρόκειται, ακριβώς τι θέλουν και τι τους χρειάζεται. Επίσης, όταν μιλάμε για τα ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να έχουμε συνεχώς κατά νου τη δυνατότητα σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, την προσφορά καθολικών υπηρεσιών και φοβούμεθα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα σωστά εργαλεία για να υποστηρίξουμε αυτές τις ε, ε, προσπάθειες. Οι υποδομές δημιουργούνται με δημόσιο χρήμα. Εκεί από εκεί αυτά ο χρήστης συνεχίζει να πληρώνει ε, στον ιδιώτη που έστησε την υποδομή αν θέλετε αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει ε, και όμως το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε κάποιες χώρες επίσης θα πρέπει επίσης θα πρέπει να δούμε ότι ε, τα ευρυζωνικά δίκτυα ε, παρέχουν υπηρεσίες που εξυπηρετούν ανάγκες πολλών και διαφόρων και του ιδιώτη χρήστη και του δημόσιου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών αρχών και Αν δείτε τώρα όσον αφορά τη χρηματοδότηση τα στοιχεία που υπάρχουν θα δείτε ότι είναι τελείως διαφορετική αν η αύξηση των κονδυλίων αυτών ή η κάλυψη των κονδυλίων αυτών α, στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούμε για την κατεύθυνση τη ευρυζωνικότητα και τη στρατηγική και θα ήθελα να κάνω τι εξή παρατηρήσει. Όταν συζητάμε την χρηματοδότηση θα πρέπει να είμαστε ακόμη σαφέστεροι και να πούμε ότι είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα του Ταμείου συνοχή και των Περιφερειακών Ταμείων, να διασφαλίσουν δηλαδή ότι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή ταχύτητα και εδώ θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις όταν δεν είναι δυνατόν να έχουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Συμφωνώ με την κυρία Βαλεάν που είπε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ιδιωτική επένδυση όσο είναι εμπορικά διαθέσιμη και από την εμπειρία μας ξέρουμε ότι χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά μπορεί να χρειαζόμαστε ακόμη υψηλότερη δυνατότητα και ακόμη υψηλότερη ταχύτητα και κάλυψη. Σε τέτοιες περιπτώσεις ε, είναι μια καλή περίπτωση στην οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε το Ταμείο Συνοχής και το Περιφερειακό Ταμείο που έχουν στόχους ε, που συνάδουν προς ε, τους στόχους της ευρυζωνικότητας. Δεύτερον, όταν συζητάμε την ευρυζωνικότητα, συνήθως μιλάμε για τις σταθερές γραμμές, οπτικές ίνες ή ε, ευρυζωνικό δίκτυο. Από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι, ότι συνδέονται αυτά. Όσοι χρησιμοποιείτε εφαρμογές ασύρματες εδώ, χρησιμοποιείτε τις ασύρματες επιλογές και παράλληλα χρησιμοποιείτε και τη σταθερή γραμμή. Και όταν βρίσκεστε έξω στην πόλη και χρησιμοποιείτε το κινητό ίντερνετ, είναι κινητό ίντερνετ μέχρι να φτάσει στην σταθερή γραμμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ε, είναι πάρα πολύ γρήγορα όσον αφορά το κινητό ίντερνετ. Οι εκτιμήσεις μας από πέρυσι μέχρι το 2014 θα μας έδειχναν μια τεράστια αύξηση. Είναι πολύ ταχεία η αύξηση. Μπορεί να έχουμε πολλαπλασιασμό επί 25-27%. Και αυτά που συζητάμε εδώ μπορεί να είναι πράγματα που ξεκινάνε από το 2013-2014 που θα αυξάνονται με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα. Και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, για τις νέες υπηρεσίες που μπορεί να προκύψουν γύρω από τις τηλεπικοινωνίες, γιατί αναπτύσσονται πολλές υπηρεσίες από ευρωπαϊκά Google και Yahoo μέχρι όλες τις εφαρμογές ε, και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα αλλά και για την ε, συνήθη παραδοσιακή οικονομία. Η βασική πρόκληση για την ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι να έχουμε αύξηση της παραγωγικότητας ε, που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την, ε, το δυναμικό αυτό που συζητάμε εδώ. Και γι' αυτό τονίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλη αποφασιστικότητα και να ανοίξουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ταχύτητα του ευρυζωνικού δικτύου. Μερικές φορές μου κάνει εντύπωση όταν μιλάμε για 100 Mbps, 2020 κλπ. Στην Νότια Κορέα ξεχνάμε ότι για το μεγάλο κομμάτι των οικοκυριών ε, έχουμε ανοιχτά χιλιάδες Mbps. Και στις ΗΠΑ Πολιτείες ε, επίσης έχουν πολύ φιλόδοξους στόχους. Για να μην συζητήσουμε καν το τι θα γίνει στην Κίνα. Και το λέω διότι μερικές φορές, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι προγραμματίζουμε τη θέση μας ως ε, υπαριθμόν τρία στο παγκόσμιο ανταγωνισμό στο μέλλον. Και ε, φοβούμαι ότι θα τα καταφέρουμε να είμαστε και νούμερο τρία, αν αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε. Όταν μιλάμε λοιπόν για την ευρυζωνικότητα, να είστε ακόμη περισσότερο τολμηροί. και όχι μόνο τα 800 MHz, ε, να στοχεύουμε ακόμη παραπάνω γιατί θα αυξηθεί η κίνηση ακόμη περισσότερο και θα πρέπει να απελευθερώσουμε και άλλα τμήματα ε, του φάσματος. Υπάρχουν οι υπηρεσίες ε, τηλεόραση και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και πρέπει να ανοίξουμε ακόμη και να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα τμήματα του, του φάσματος όσο το δυνατόν καλύτερα και αποδοτικότερα. Σεβόμενοι τις πολιτισμικές διαφορές, λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι πολιτισμικές διαφορές συνεισφέρουν ε, στην ανάπτυξη. Το 70% της κίνησης στο κινητό ίντερνετ είναι βίντεο και όχι μόνο YouTube, αλλά και με σοβαρό πολιτιστικό περιεχόμενο. Άρα και ο πολιτισμός εδώ θα βοηθήσει. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν και να προσδιορίζουμε εμείς το μέλλον των συζητήσεων αυτών για να μην είμαστε νούμερο 3 ή νούμερο 4, αλλά να αναλάβουμε τη δέσμευση ότι θέλουμε να γίνουμε νούμερο 1. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δύο λεπτά μας έχουν μείνει. Και θα ήθελε το λόγο και η συνάδελφος Τικά, αλλά πάρα πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία και στην εισηγήτρια να μιλήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Τζαβέλα για το έγγραφο που μας ε, έχει παρουσιάσει. Συζητάμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για την ανακοίνωση της Επιτροπής. Ε, δυστυχώς, αν το 2008, όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση, ε, είχε δεσμευτεί η Επιτροπή ότι θα προσφέρει 100% κάλυψη ευρυζωνικότητας μέχρι τα τέλη του 2010. Επειδή δεν καταφέραμε να το κάνουμε, με κανονισμό δεν το προωθήσαμε και τελικά δεν υλοποιήθηκε δεσμεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2013 να το κάνει. Ελπίζω ότι μετά την έκθεση αυτή θα αντιδράσει η Επιτροπή με ένα έγγραφο που θα τη δεσμεύει να φτάσει πραγματικά το στόχο αυτό. Νομίζω ότι έχει σημασία να συζητήσουμε και το θέμα της ε, συμμετοχής όλων των πολιτών στην ε, ψηφιακή εποχή και θα πρέπει να καλύπτει το ευρυζωνικό δίκτυο και τις πιο φτωχές περιοχές. Πρέπει να μιλάμε για την ευρυζωνικότητα ως ένα είδος καθολικής υπηρεσίας. Όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτού είδους τις υπηρεσίες. Και τέλος, θα ήθελα να αναφέρεται στην έκθεση η ενδιάμεση αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών, ούτω ώστε να έχουμε την εγγύηση ότι η κάλυψη 100% μέχρι το 2013 θα είναι κάτι που πραγματικά θα υλοποιηθεί. Αυτά και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τζαβέλα και πάλι. Δεν ξέρω αν θέλει η Επιτροπή να πει κάτι. Αν δεν θέλετε. Ελπίζω να μην έχετε μισή ώρα συνεισφορά. Απλώ θέλουμε να συγχαρούμε την εισηγήτρια και να πούμε ότι χαιρετίζουμε την έκθεση. Τίποτα άλλο, κύριε Πρόεδρε. Μία από τι καλύτερε παρεμβάσει που ακούσαμε σήμερα. Κυρία Τζαβέλα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους που πήραν το λόγο. Ήταν πολύ επικοδομητική και ε, συζήτηση και χάρηκα πολύ. Οι ιδέες ήταν πολύ σημαντικές για, μα, για μένα και με εμπνέουν και με υποκινούν να κάνω μια καλή έκθεση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πράγματι σημείωσα, σημειώσαμε όλα αυτά που ελέγχθησαν εδώ. Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας και έτσι θα καταλήξουμε σε μια έκθεση η οποία θα είναι ανοιχτή προς το μέλλον. Συμφωνούμε όλοι θα ότι εδώ πρόκειται για ένα από, το πιο, από τους πιο σημαντικούς τομείς στην Ευρώπη. Ένα σχόλιο όμως έχω να κάνω. Να σας πω ότι εγώ επιφυλάχθηκα λιγάκι στο να ανα, το να βάλω ακόμη να κάνω την έκθεση ακόμη πιο φιλόδοξη γιατί ε, δεν ήμουν σίγουρη για τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα ήταν διαθέσιμα. Εν πάση περιπτώσει όμως όλα αυτά που ελέγχθησαν τα σημειώσαμε ήταν πολύτιμα για μας η συζήτηση ήταν πάρα πολύ καλή και κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ. Θα βελτιωθεί λοιπόν η έκθεσή μας για την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος για τις τελικές σας παρατηρήσεις. Σας εύχομαι καλή δουλειά για σήμερα. Απλώς καλό βράδυ. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί. Γεια σας.